αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Και καλωσορίζω τα μέλη της Επιτροπής Ενεργείας και Μεταφορών της Γερουσίας της Ρουμανίας. Είναι μαζί μας. και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γερουσίας για Ενέργεια και Μεταφορές. Είναι εδώ. Λοιπόν, η Επιτροπή μας ε, μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών ήταν μαζί μία και το ε, ήτρε από τις μεταφορές. Μας, λείπει, μας λείπουν οι μεταφορές αλλά παρόλα αυτά έχουμε πολλές δραστηριότητε και μία από τις σημαντικότερες είναι οι επενδυτικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, στις υποδομές, στη βιομηχανία και ο βασικός υπεύθυνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά σήμερα είναι ο αντιπρόεδρος ο κύριος Γιούρκι Κατάινεν, πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, είναι μαζί μας Μιλάμε για το διαφρομένο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσία σας εδώ. Πολύ συχνά ερχόσαστε και το θαυμάζουμε. Είστε Αντιπρόεδρος υπεύθυνο για την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Με αυτή τη σειρά και όχι την αντίστροφη. Πάντα από ανταγωνιστικότητα πρέπει να ξεκινάμε για να καταλήξουμε σε περισσότερες απασχόλησεις. I, I Προσπάθησα να αλλάξω κάπως το χαρτοφυλάκι του και περιεχόμενο με διαφορετική σειρά όπως βλέπετε ακολούθησα. Ο κύριος Κατάινεν συχνά επισκέπτεται την Επιτροπή μας, την Ήτρε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους σας ότι η Ήτρε είχε συμμετάσχει κατά πολύ στην υιοθέτηση ε, ε, του κανονισμού για το ΕΦΣΥ. Η κυρία Βαν Μπρέντ, η συγκήτρια, είναι μαζί μας. And, ε, το άρθρο 54 είναι ειδική για την πηγή χρηματοδοτήσεως και τους τομείς επενδύσεων είναι η Επιτροπή μας και θέλουμε να παρακολουθήσουμε εκ του στην στην εφαρμογή ε, του μέσου αυτού. Κύριε Αντιπρόεδρε, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάντα χαρά να είμαι μαζί σας. Θα καλύψω πολλά ζητήματα του προγράμματος εργασίας ε, που σχετίζονται με το δικό σας έργο στην Επιτροπή αυτή εδώ. Αλλά πριν πω στην ουσία, πρέπει να πω ότι μου αρέσει αυτός ο διαρθρωμένος ε, τρόπος ε, συζήτησης ε, ώστε να ακούμε και από το Κοινοβουλίο τι αλλαγές θα πρέπει να κάνουμε του χρόνου, ειδικότερα πριν από το την ε, έναρξη της προετοιμασίας του προγράμματος εργασιών του επόμενου έτους. Οπότε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Ας ξεκινήσουμε από το φλέγον θέμα τη σημερινή ημέρα το χάλιβα. Όπως γνωρίζετε η χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δύσκολες εποχές και έχει γίνει έκκληση για δράση τόσο από τις βιομηχανίες όσο και από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν ε, εδώ και έξι μήνες προσπαθεί να μελετήσει την αντιμετώπιση του ζητήματος ε, στο Συμβούλιο και σε μια διάσκεψη τον περασμένο μήνα. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε τι προβλέπουμε με αυτό το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη 37 διαφορετικά μέτρα για την χαλιβουργία και 16 μέτρα που αφορούν τις εισαγωγές χάλιβα από την Κίνα. Ε, και όσον αφορά τις διαδικασίες και τα επίπεδα τελών. Τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασίζονται στη συμμετοχή των κρατών μελών σε ε, στάδια κλειδί της έρευνας. Ε, πραγματοποιεί εννέα έρευνες η Κομισιόν. Θέλει να κάνει μια πλήρη ανάλυση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζοντας για παράδειγμα τα συμφέροντα των χρηστών και εφαρμόζοντας τον κανόνα του χαμηλότερου τέλους. Το interest test Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή η Κομισιόν ξεκινά μια έρευνα βάσει της απειλής ε, τραυματισμού. Είναι ένα νέο μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε τώρα. Ε, Ουσιαστικά δεν περιμέναμε να υπάρξει τέτοιος τραυματισμός, αλλά, να, ε, αλλά ε, λειτουργούμε βάσει απειλής. Και προσπαθούμε να απελύνουμε την κατάσταση πριν εφαρμοστούν ε, προσωρινά μέτρα, ώστε να εφαρμόσει η Κομισιόν τέλη αντι πριν από την υιοθέτηση των μέτρων. Κάνουμε πράγματα που δεν χρειάζονται νομοθετικέ αλλαγές. Μειώνουμε τη διαδικασία κατά ένα μήνα από το μέσο όρο των 9 μηνών στους 8. Θα αυξήσουμε τη χρήση της γραπτής διαβούλευσης. Κατά τη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Εμπορίου πριν υιοθετήσουμε προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά μέτρα επίσης μπορούν να επιβληθούν από την Κομισιόν μετά από ενημέρωση των κρατών μελών σε περίπτωση ε, έκτακτων αναγκών. Η Κομισιόν θα βελτιώσει περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες μέσω μιας αυστηρής προσέγγισης ώστε να ασχοληθεί με ε, παρατάσεις, με απαντήσεις σε ερωτήσεις, ε, ομαδοποιώντας τα αιτήματα. Επίσης, θα θέλαμε οι συνομοθέτες, δηλαδή το Συμβούλιο, κυρίως να αναλάβουν τις ευθύνες τους κατά τον εξυγχρονισμό των ε, μέσων ε, υπεράσπισης του εμπορίου. Το πακέτο του Απριλίου 2013 αποτελεί από μία ανακοίνωση, μία πρόταση ε, κανονισμού με σχέδια κατευθυντήριων γραμμών μη δεσμευτικών και κάποιους στόχους αυξημένη διαφάνεια και προβλεψιμότητα, καταπολέμηση κατά των αντιμέτρων, καλύτερη αποτελεσματικότητα και επιβολή, ευκολότερη διαδικασία συνεργασίας, βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης και κωδικοποίηση ορισμένων πρακτικών στην νομοθεσία. Ενώ αρχικά δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά μέσα υπεράσπιση του εμπορίου, ο κανονισμός εξυγχρονισμού προσφέρει ε, τη δυνατότητα τροπολογιών κατά την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία. Ε, αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και στη Χαλιβουργία και όχι μόνο σε περιπτώσει διαστρέβλωση τη αγορά ε, πρώτων υλών. Αυτό είναι δυνατόν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και επίση θα πρέπει να οριστεί καλύτερα ε, το κέρδος στόχος για τον υπολογισμό του ε, περιθωρίου ζημίας ώστε να απαλληφθούν οι ζημιές. Οι ζημίες τι θα μπορούσαμε να κάνουμε επιπλέον το οποίο απαιτεί νομοθετικές αλλαγές. Ε, και θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της πρότασης εξυγχρονισμού του μέσου υπεραυσής του εμπορίου, μειώνοντας τη διαδικασία κατά δύο επιπλέον μήνες σε 7 ή 6 μήνες μέσω αλλαγών στους κανονισμούς ε, κατά των επιχορηγήσεων και anti-dumping ε, προθεσμίες ε, θα μπορούσαν να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές. Επίσης η διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προστευθεί χωρίς να επιτρέπει η διαδικασία ε, έφεση στα τελικά, έσταση στα τελικά στάδια. Τέλος, ε, επιτήρηση εκ των προτέρων ε, των, της χαλιβουργίας, μέτρα που προβλέπονται στο, και βασίζονται σε ένα σύστημα αδειοδότησης των εισαγωγών. Μπορούν να εισαχθούν όταν υπάρχει απειλή από εισαγωγές για τους εγχώριους παραγωγούς. Αυτά όμως κυρίες και κύριοι είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι της δράσης το εμπόριο δεν εξηγεί όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανοί μας αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία μας, να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα ενδιαφέρονται να μάθουν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, οπότε σας ενθαρρύνω να το διαβάσετε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα. Τώρα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του 2016, η υλοποίηση βρίσκεται σε καλό δρόμο, η αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων παραμένουν στην ατζέντα. Το ΕΦΣΥ λειτουργεί κανονικά και τώρα βελτιώνουμε το επενδυτικό περιβάλλον και ε, αποκομίζουμε τα ωφέλη των ευκαιριών. Θα σας ενημερώσω γι' αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο στόχος είναι να δώσουμε μια όθηση στην ενιαία αγορά, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αέροντας τα ε, διάφορα εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Μια σειρά πρωτοβουλίων βρίσκονται σε προετοιμασία όπως διατυπώνεται στη στρατηγική μας για την ενιαία αγορά το τελευταίο Οκτωβρίου του περασμένου Οκτωβρίου. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το, το πιο σημαντικό κομμάτι του επενδυτικού σχεδίου, ο τρίτος πυλώνας έτσι ονομάζεται. Επίσης παρακολουθούμε την εξέλιξη της ψηφιακής ε, και ενεργειακής μας στρατηγικής. Ε, αναφέραμε τα δικαιώματα και το copyright ε, τον περασμένο Δεκέμβριο με κάποια μέτρα που θα εφαρμοστούν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές καθώς και η αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των καταναλωτών. Σε όλους αυτούς τους τομείς η προστασία των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα κομμάτι όλων των προσπαθειών μας να αξιοποιήσουμε τις πλήρες ε, δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Παρακολουθούμε τις πέντε εκθέσεις ε, προεδριών για την ε, EFU. Ναι. Ξεκινάμε μια διαβούλευση για το, ε, ξεκινήσαμε μια διαβούλευση για τα ε, κοινωνικά δικαιώματα την περασμένη εβδομάδα και προετοιμάζουμε μια νέα ατζέντα δεξιοτήτων για το Μάιο. Έχοντα επενδύσει σημαντικέ προσπάθειε ε, για τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού, τώρα πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Προωθούμε το σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία του περασμένου Δεκεμβρίου, προσπαθώντα να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο ε, μέλλον για την Ευρώπη βάσει της στρατηγικής 2020 και τους ε, στόχους αηφόρου ανάπτυξης. Να πω δύο λόγια για το κοινό μας εμβληματικό έργο της ε, στρατηγικής για την Ευρώπη. Αρχίζουν και αποφέρουν αποτελέσματα. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 54 έργα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 54 λοιπόν έργα, 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και άλλα έργα θα συνεχίσουν να επιλεγόνται. Από τα μισά από αυτά τα έργα υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και άλλες μεθόδους μείωσης των εκπομπών. Ε, περιλαμβάνουν επίσης έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορές, υποδομές, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο έχει υπογράψει πάνω από 150 συμφωνίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολική χρηματοδότηση ύψους 3,4 δις ευρώ. 125.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν. Όλες αυτές θα οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις περίπου 76 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρώτων 7 μηνών. 76 δισεκατομμύρια. 22 κράτη-μέλη έχουν αποφεληθεί από το ΕΦΣΥ και μικρές οικονομίες όπως η Σλοβενία, η Εσθονία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν ήδη να ζητήσουν τεχνική αρρωγή από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδύσεων, Συμβουλευτικό Κόμβο Επενδύσεων. Αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσουμε και την πύλη επενδύσεων για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ε, ώστε να διαφημίζουν σε πιθανούς επενδυτές τα προϊόντα τους. Ε, κάτι που είχε συζητηθεί από τον τομέα. Τέλος, ε, η Επιτροπή επιδιώκει μια φιλόδοξη ατζέντα άρσης συγκεκριμένων ρυθμιστικών και διοικητικών εμποδίων για τις επενδύσεις και για τη δημιουργία ενός καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Ψάχνουμε με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χώρες και 26 Νοεμβρίου πέρυσι υιοθετήσαμε μια νέα προσέγγιση που αφορά συγκεκριμένα δελτία για χώρες ε, με αναφορά στα εμπόδια προς επενδύσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη η Κομισιόν έχει ξεκινήσει την Ένωση Κεφαλαιογορών, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την στρατηγική ενιαία αγορά. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Στις 27 Φεβρουαρίου, στις 22 Φεβρουαρίου, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσαν ε, ένα έγγραφο που θα βοηθήσει τις ε, τοπικές αρχές και τους διάφορους φορείς να αξιοποιήσουν το συνδυασμό των κονδυλίων Εύση και ΕΣΥ. Αυτά τα δύο μέσα έχουν, αποφασιστεί, έχουν σχεδιαστεί με συμπληρωματικό τρόπο. Ενισχύουν το ένα το άλλο. Να πω δύο λόγια για την ε, άλλη μου βασική ευθύνη για φέτος, την κυκλική οικονομία. Αυτή είναι η βασική συνεισφόρα στις προτεραιότητες που θέτουμε και το θεματολόγιο για ανάπτυξη και απασχόληση και συνδέεται στενά με την πολιτική ενέργεια και το κλίμα και σε μια εποχή προβλημάτων και δεσμεύσεων για την αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο και το ευρύτερο πρόγραμμα για το 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη που θέτει και από τον ΙΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο που θα γεννηθούμε Η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλλει κατά πολύ σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Το πακέτο αποφασίστηκε με ευκαιρίες επιχειρηματικές που θα είναι βιώσιμες σαν στόχο. Η κυρκική οικονομία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο στις λύσεις της πράσινης και την πράσινη τεχνολογία. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις πηγές μας, να μειώσουμε την εξάρτησή μας σε σπανίζοντα σε σπανίζουσες πρώτες ύλες τότε μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση. Τα νέα μοντέλα στην κυκλική οικονομία μπορούν να παίξουν έναν μεγαλύτερο ρόλο. Εντό του ορίζοντα 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη επενδύει πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα επιδείξει για ανανεώσιμα σε μία διετία. Στα πέστη κυκλική οικονομία εστιαζόμεθα ε, στι επενδύσει για βιώσιμε υποδομέ που θα πρέπει να φτιαχτούν στα πλαίσια των Ιθωτικών ταμείων και του ΕΦΣΥ και κάνουμε και άλλε δοκιμέ. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τι Εθνικέ Τράπεζε για να προωθήσουμε τι επενδύσει στην κυκλική οικονομία. Επίση, το ΕΦΣΥ εντοπίζει την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων σαν βασικό στόχο. Πέρα από τη χρηματοδότηση παραδοσιακή, δημιουργεί δυνατότητε για να προωθήσουμε προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και υποστηρίξουμε τη μεταμόρφωση προ την κυκλική οικονομία που χρησιμοποιεί ε, λίγα ορυκτά καύσιμα. Ε, κύριε Πρόεδρε, να πω και μερικά λόγια κλείνοντας ε, για τον ορίζοντα 2020. Ε, όπως προανέφερα, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όμως γνωρίζουμε ότι η έρευνα και, και επενδύσεις για την έρευνα είναι το μέλλον είναι ακρογωνίως λίθος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προωθήσει την έρευνα για την ανάπτυξη και, την, και της απασχόλησης. Ο Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα το ερευνητικό 77 δις έχουμε διαθώσει, 2,2 δισεκατομμύρια πήραμε από τα χρήματα για να δημιουργήσουμε το ΕΦΣΥ και αυτό μας έδειξε ήδη μετά από μερικούς μήνες ότι το ΕΦΣΥ θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την καινοτομία πολύ παραπάνω από αυτά που θα επέδιδαν τα 2,2 δις. Τα δύο τρίτα τα προγράμματα του ΕΦΣΙ αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Ο ορίζοντας 2020 πετυχαίνει τους στόχους. 7.200 συμφωνίες έχουμε συνάψει για χορηγίες με συνεισφορά 12,6 δις ευρώ σε 31.000 συμμετέχοντες. 7.200 συμφωνίες για χορηγίες, 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ για 31.000 φορείς που συμμετέχουν. Πάνω από 1.300 συμφωνίες για χορηγίες με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ερευνών. Λοιπόν, η προετοιμασία των προγραμμάτων έλαβε υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ειδικέ μελέτε, αποτελέσματα διαβουλεύσεων σε εμπλεκομένους φορείς και προτεραιότητες Ευρωπαϊκή Ενώσεω, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία που έχει σωστό στόχο και κλίμακα, να δώσουμε προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή επίση. Στο πρόγραμμα εργασιών των παρών, 670 εκατομμύρια ευρώ για τη βιομηχανία, στην κυκλική οικονομία, στην βιομηχανία ή 139 εκατομμύρια ευρώ για το διαδίκτυο των αντικειμένων, των πραγμάτων. Βρήκαμε επενδυτικέ ευκαιρίε επί διετία, με ένα πλουστευμένο πρόγραμμα εργασιών. Οπότε η κοινότητα έρευνα και ανάπτυξη έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα. Ορίζον 2020 είναι πολύ ελκυστικό πρόγραμμα. 84.000 προτάσει υπευλήθησαν μέχρι τώρα. Ζητούν 246 δις ευρώ. Δις σας λέω και αυτά τα μέτρα ε, είναι πιο προσβάσιμα από ποτέ. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Horizon 2020 ε, θα κάνει μια αποτίμηση. Θα σταθμίσει και θα βελτιώσει την υλοποίηση του ορίζοντα 2020 για την εναπομένουσα περίοδο προγραμματισμού και χρηματοδοτήσεως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομιών έχει ζητήσει υποβολή ιδεών για να μπορεί το Συμβούλιο να στηρίξει τους πολλά υποσχόμενους καινοτόμους φορείς. Ε, θα έχουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ψηφιακό κόσμο και θέλουμε να ακολουθήσουν τις δέουσες στρατηγικές οι χώρες που θα διευκολύνουν την προσέγγιση μας στην ψηφιακή αγορά. Και θέλουμε να δούμε και πώς τα προγράμματα πλαίσια επηρεάζουν τις εξελίξεις και πόσο μπορούμε να δημοσιεύουμε τι έρευνε και τα στοιχεία όσον αφορά την έρευνα, να λάβουμε υπόψη τα θέματα ασφαλείας και να προσθέσουμε τα διάφορα μέτρα που ε, ομολογούμε. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κύριε Πρόεδρε, αλλά βλέπετε έχετε ευρύτατο το θεματολόγιο. Προσπάθησα να καλύψω τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεμάτων που σα ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, λέει ο κ. Μπούζεκ, και για την οριζόντια προσέγγισή σα. Σα ευχαριστώ. Με επί τρόπου συνεργάζεστε από ό,τι θυμάμαι. Άρα το χαρτοφυλάκι σας είναι ευρύτατο. Συνάδελφοι, που θα πάρετε το λόγο εσείς που εκπροσωπείτε πολιτικές ομάδες, παρακαλώ, όχι πάνω από δύο λεπτά και οι άλλοι συνάδελφοι ένα λεπτό, διότι μας λείπει ο χρόνος. Και έχουμε μακροσκελή κατάλογο ομιλητών. Αυτό βλέπω μπροστά μου. Ο κύριος Έλερ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Um, Χαίρομαι που σας βλέπω, Επίτροπε. Ελπίζω να μην είναι μόνο διαρθρωμένος διάλογος, αλλά και επικοδομητικός. Το πρόβλημα με το δίλεπτο είναι πώς να, τι να πεις σε δύο λεπτά. Για το χάλιβα έχω απλή ερώτηση. Εσείς ανησυχείτε λέτε για τους όρους ε, των εμπορικών συναλλαγών μας και την ανταγωνιστικότητα που έχουμε με την Κίνα και το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Ε, οι πάντες έχουν εξαγριωθεί, τα συνδικάτα, η χαλιβουργία στη χώρα μου. Ε, σου λένε θέλετε να μας πετάξετε έξω από την αγορά. Και το κόστος για την εκλογική μου περιφέρεια για τη χαλιβουργία για ένα νέο σύστημα ETS θα ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν πια επενδύσεις στην εκλογική μου περιφέρεια. Και έχει γίνει ένα out. Οι νέες επενδύσεις δεν θα έρθουν στην Ευρώπη πια και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στην περιοχή από το Σαλτσκίτερ και λοιπά, έχουν φύγει εταιρείε πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι θα γίνει λοιπόν τώρα με αυτό, ε, με τον αθέμητο ανταγωνισμό, το αθέμητο εμπόριο και το επιπλέον ε, βάρος από το σύστημα εμπορίας εκπομπών για τον ορίζοντα 2020 και το Ταμείο ε, Στατηγικών Επενδύσεων το ΕΦΣΥ. Χαίρομαι αυτά που κάνετε για τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα το είναι φίν. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως εκεί που κατά την άποψή μου είναι λίγο πρόβλημα και αυτό είναι τα κριτήρια για τις βιομηχανίες ε, της δημιουργίας. Είναι μεγαλύτερη από τη φαρμακοβιομηχανία, από το αυτοκίνητο βιομηχανία από τη χαλιβουργία. Η δημιουργική κλάδη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό στην Ευρώπη. Uh, Ευχαριστώ ε, κυρία Βαν Μπρέντ, εξ των σοσιαλιστών. Ε, Ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε στα διαφορετικά αυτά θέματα. Αν υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή σε αυτό είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία μας. Αυτό ξέρουμε όλοι και να επενδύσουμε στην οικονομία μας. Και ή θα είναι βιώσιμη ή δεν θα υπάρχει. Έτσι πρέπει να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Εν αυτή τη ενία το Ευρωπαϊκό Σταμείο Στατηγικών Επενδύσεων δεν θα επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές που θα θέλαμε, τις μεγάλες, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο τουλάχιστον να μας βοηθήσει να κινηθούν προς τα εκεί. Και αυτό είναι το βασικό σημείο που προωθούσε αυτή η Επιτροπή όταν εισήλθε στις συζητήσεις μέσω τροπολογιών και εκθέσεων και στις συζητήσεις με τα τρία θεσμικά όργανα που διεξήχθησαν για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Θέλουμε βιωσιμότητα, όχι να είναι αυτοσκοπός οι επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις να χρησιμοποιούνται ούτω ώστε να αλλάξει η οικονομία. Αυτό σχετίζεται με το βασικό μου ερώτημα, οι ερωτήματα. Για μας είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να δούμε αν, κατά πόσο πετύχαμε, αν πλησιάζουμε το στόχο. Υπάρχουν πολλά έργα και προγράμματα στον κατάλογο, την πρώτη διαλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα προγράμματα, πολύ δύσκολο για μας να αξιολογήσουμε φερρυπίν το σύστημα των πίνακα βαθμολόγησης του ΕΦΣΥ. Πώς χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται εκ των προτέρων. Μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα περί αυτού. Και το κοινό μπορούμε να δούμε πώς γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων και πώς βαθμολογούνται στον πίνακα βαθμολόγησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, η ενεργειακή απόδοση, πολύ σημαντικό θέμα και για αυτή την Επιτροπή και σχετίζεται με πολύ μικρά έργα και προγράμματα που είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι πιο εύκολο να επενδύσει κανείς σε μεγάλα έργα, πολύ δύσκολο είναι να δρομολογηθούν αυτά τα μικρά προγράμματα στα κράτη-μέλη. Δεύτερη ερώτηση. Άρα πώς λειτουργούν τα πράγματα, οι πλατφόρμες πώς λειτουργούν, η συνεργασία πώς οργανώνεται. Είναι πολύ καλή η πρόταση στη, Γαλλία για την απόδοση της θέρμανσης στα κτίρια, τις κατοικίες. Πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει σε ένα τέταρτο να φύγω, αλλά ο βοηθός μου είναι εδώ για να ακούσει τις ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ, κυρία μου. Κυρία Κάλλας, εξ του Άλντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα κυρία σημεία που αναφέρατε. Όπως όλοι γνωρίζουμε για τις θέσεις εργασίας και για την ανάπτυξη για, του είδους, για τις θέσεις εργασίας που θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε την έρευνα και την καινοτομία. Οπότε η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Μπροστά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεταναστευτική κρίση και όλα τα υπόλοιπα, εμφανίζονται και διάφορα επιπλέον κόστη. Πώ είστε βέβαια, τι εγγύηση υπάρχει ότι δεν φεύγουν αυτά τα λεφτά από τον προπολογισμό της έρευνας και της κοινοτομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μαραγκάλ, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ για αυτή την ενημέρωση. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε. Ε, μερικές ερωτήσεις. Ε, ε, κάποιες γενικές παρατηρήσεις καταρχάς. Ε, όσον αφορά τη λειτουργία του κόμβου, ε, ε επιτυχάνει τους στόχους, εκπληρώνει τις προσδοκίες, ε, πώς χρησιμοποιείται η πύλη, ε, πώς πάει. Χρησιμοποιείται. Και μετά, όπως μόλις υπόθηκε, Πώς πάει ο πίνακας βαθμολόγησης. Λοιπόν, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Κάποια παραδείγματα, κάποια παρατηρήσεις, δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα σημεία, αλλά για κάποια μπορώ. Ε, θα σας πω κάποια πράγματα που αφορούν την Ισπανία τώρα για τις νέες τεχνολογίες ε, ε, ε, μιλώ για τα φίλτρα ελέγχου ε, που πρέπει να περάσουν τα πράγματα έχουν περάσει από αυτό με τα τρία έργα αυτοκινητοδρόμων ένα στις κατοχώρες, ένα στη Σλοβακία και ένα στη Γερμανία ένα 500 εκατομμυρίων στη Σλοβακία 100 εκατομμυρίων στις κατοχώρες όλα αυτά είναι χρήματα για αυτοκινητοδρόμους Αυτά πληρούν τα κριτηριά σας, τα κριτηριά μας όταν κοιτάμε τον, την προσθετικότητα του κανονισμού ΕΦΣΙ. Υπό την ίδια έννοια, επενδύσεις σε δηληστήρια στην Ιταλία, 13 εκατομμύρια από το ΕΦΣΙ. και αυτό έχουμε και την ισπανική περίπτωση με τα δύο πλοία που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΦΣΙ επίσης Μιλάμε για, μια, για πολλά παραδείγματα που μας δείχνουν πώς πραγματικά εφαρμόζονται τα κριτήρια του ΕΦΣΥ. Τώρα μια γενική ερώτηση. Ποιο είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται με αυτά τα 70 δις που αναφέρατε. Είναι 15 πλάσιο το αποτέλεσμα. Πόσο είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφα. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δουν νέα κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες να δώσουν όθηση στην πραγματική οικονομία. Γιατί μόναχα έτσι μπορεί να υπάρξει διέξοδος από την κρίση και την ύφηση και να υπάρξει πραγματικό όφελος προς όφελος της κοινωνίας και των λαών. Δυστυχώ όμω αντί αυτού η Κομισιόν επικεντρώνεται στη διασφάλιση των εγγύσεων ώστε να μειώσει το ρίσκο των ιδιωτικών επενδύσεων των μεγάλων εταιριών. Είναι προβληματικό το γεγονό ότι παρόλο που η Κομισιόν υποσχέθηκε να δώσει κονδύλια για επενδύσει, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να περικόπτει ε, κονδύλια από της τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω τα 16 δισεκατομμύρια από το στρατηγικό σχέδιο επένδυση αρκετά προέρχονται από περικοπέ από το πρόγραμμα Horizon, από το πρόγραμμα Συνδέοντα στην Ευρώπη. Και δυστυχώ γίνεται ξεκάθαρο πω τα ε, τα κονδύλια αυτά πηγαίνουν κυρίω σε ανεπτυγμένα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στα κράτη των οποίων η οικονομία έχει διαλυθεί λόγω των μνημονιακών νοφιλεύθερων πολιτικών τη σκληρή λιτότητα. Και θα φέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Για παράδειγμα, πώ δικαιολογείται το γεγονό ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 η Ελλάδα και η Κύπρος απουσιάζουν εντελώ από το επενδυτικό σχέδιο τη Κομισιό. Γιατί δεν έχει περιληφθεί κανένα πρόγραμμα ούτε στα 42 προγράμματα ε, των υποδομών και τη καινοτομία, αλλά ούτε και στα 84 προγράμματα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αυτέ τι δύο χώρε που υποφέρουν με κρίση και ύφεση. Και ακριβώ το ερώτημα μου, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι πώ προτίθεται η Κομισιόν να στηρίξει ακριβώ αυτά τα κράτη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανάπτυξη λόγω και των μνημονιακών μέτρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, e Ευχαριστούμε πολύ εκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σκέψεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός. Πρώτον, κύριε Αντιπρόεδρε, αναφέρατε τα μέτρα αντι-dumping. Εγώ να σας ρωτήσω, δεδομένου ότι η Κομισιόν φαίνεται να κινείται προς την εκχώρηση της οικονομίας αγοράς ε, στην Κίνα, όπου πλέον αυτά τα μέτρα δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν. Τώρα το ευχόμαστε να ξεμπλοκάρει η έκθεση των μέσων ε, υπεράσπισης του εμπορίου. Εντάξει το πιστεύω, αλλά ως επιχειρηματίας εγώ τώρα ε, δεν θα έκανα ε, δουλειές βάσει ευχολογίου. Δεύτερο, πριν από λιγότερο από ένα χρόνο κόψαμε κονδύλια από το ορίζοντα 2020 για να χρηματοδοτήσουμε το ΕΦΣΙ που θα επέστρεφε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα στα τέσσερα σχέδια σήμερα του ορίζοντα 2020 ε, κατευθύνεται προς το μέσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά έχουμε χρηματοδοτήσει μόνο τα μισάρια στην περίπτωση της Ιταλίας, διότι δεν έχουμε επαρκή κονδύλια. Παρότι οι επιχειρήσεις μας ε, ε, έφεραν προγράμματα εξαιρετικά. Να σας ρωτήσω λοιπόν, αν βάζαμε μισό δις, ε, όχι μεγάλα ποσά όπως αυτά που είπατε εσείς, μισό δισεκατομμύριο στο Ταμείο Εύση για το κομμάτι του ορίζοντα 2020, ειδικά για το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αύριο το πρωί, όχι σε ένα χρόνο, θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε έργα μικρομεσαίων επιχειρήσεων αριστείας ε, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καινοτομία άμεσα στην Ήπειρό μας, δημιουργώντας αυτό το σύστημα εμπιστοσύνης που θα μπορέσει να βοηθήσει στη συνέχεια και τους εξωτερικού, να έρθουν εξωτερικοί επενδυτές στην Ήπειρό μας. Ε, τι σκέφτεστε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ έχει το λόγο εκ μέρους ομάδα της. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μου αρέσει ο τρόπος ε, με τον οποίο ξεκινήσατε το σημερινό διάλογο με το θέμα του Χάλιβα ήταν κατεπήγον θέμα επί σημαντικό χρονικό διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Χαλιβουργίας που έχει υποφέρει από πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα αφορά και το anti-dumping. Βλέπουμε 100.000 τόνους δυναμικό έχουμε όσον αφορά το χάλιβα που έρχεται από την Κίνα αυτή η ποσότητα και από τρίτες χώρες. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό και πρέπει να εξυγχρονιστούν και τα μέτρα προστασίας του εμπορίου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε ότι οι δασμοί αντι-dumping θα πρέπει να εφαρμοστούν. Κοίτα, κοιτάξτε τι, κάνει, τι κάνουν οι Αμερικανοί. Γιατί η Χαλιβουργία είναι κλασικό κλάστερ για την ανάπτυξη, την απασχόληση εκατοντάδε χιλιάδες θέσει εργασίας και στη στρατηγική 2020 με το στόχο να έχουμε 20% ε, επαναβιομηχάνηση στην Ευρώπη. Και εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε τις μεγάλες βιομηχανίες, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό γιατί αλλιώ ε, όλοι οι υπηρεσία, όλη, όλος ο κλάδος των υπηρεσιών ε, υποφέρει. Και μια που μιλάμε για τη χαλιβουργία είναι και ένα δεύτερο θέμα. Το θίξατε λίγο, ακροθυγός είναι η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα ενεργειακές τιμές, η τιμολόγηση. Το είπε και ο προλαλής σας, ε, ότι φεύγουν πολλές χαλιβουργίες και από την Αυστρία, από την εκλογική μου περιφέρεια υπάρχει μια μεγάλη χαλιβουργική που πάει στις ΗΠΑ τώρα και ε, επεκτείνεται γιατί είναι ε, χαμηλό και το κόστος εργασίας και ενέργειας και το μη μισθολογικό κόστος και πάει λέγοντας εμείς πώς μπορούμε τις μεγάλες μας εταιρείες να τις κρατάμε στην Ευρώπη ανταγωνιστικές. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα το οποίο αναφέρεται είναι η ψηφιοποίηση. Μόλις άνοιξε η έκθεση Τσέμπιτ, έκανε εγγένεια η μεγάλη έκθεση αυτή και τι γίνεται με τις τεχνολογίες blockchain για τις ε, οικονομικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και είναι σημαντικό αυτό και για το μέλλον. Τεράστιες εξοικονομήσεις μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη παντού και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Αυτά τα δύο ερωτήματα είχα και ε, αν μου επιτρέπετε ένα σύντομο για το Τραμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, μιλήσατε για τα σχέδια, ο πρόεδρος διακόπτη, για τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόθεση. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο σχετικά. Uh, λοιπόν, ε, τώρα πάμε στα μονόλεπτα. Δηλαδή πάμε πάρα πολύ, δεν έχουμε χρόνο. Ο συνάδελφος Νίκα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε για την χαλιβοργία. Ο τύπος λέει ότι είναι δειλά αυτά που προτείνεται και πολύ λίγα. Μιλάτε για μείωση των διαδικασιών ε, αντι-dumping ε, κατά δύο μήνες, μείωση της διάρκειας. Στις ΗΠΑ είναι δύο μήνες τελεία η σύνολη διάρκεια. Ε, έχουμε εδώ ένα γκρουπ από τη γερουσία της Ρουμανίας που παρευρίσκεται και παρακολουθεί τις εργασίες μας στη Ρουμανία ενδιαφέρονται για το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και 300 τόσα δις ε, του Ταμείου αυτού. 315 αν δεν απατώμε. Ε, και οι τράπεζες ενδιαφέρονται και άλλοι φορείς, αλλά ούτε ένα έργο δεν έχει εγκριθεί για τη Ρουμανία. Πώς είναι δυνατόν και πώς θα καλύψει το έλλειμμα που τη χωρίζει από τις άλλες χώρες ο κύριος Λεβαντόφσκι. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι και εκτιμώ τις προσπάθειές σας και για το Ταμείο Στρατηγικών Επενθύσεων. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το προφίλ των έργων του ΕΦΣΥ σε σχέση με τον ορίζοντα ως προς τον κίνδυνο και ποια είναι η γεωγραφική τους κατανομή. Αλλά μια γενική ε, ε, παρατήρηση στο ευχολόγιο όταν ρωτάμε τις βιομηχανίες τι θέλετε για να είστε ευτυχείς μας λένε να μειώσετε την κανονιστική ανασφάλεια να μειώσετε το άχθος αυτό μετά σου λένε για το φόρο και μετά σου λένε για τις τιμές της ενέργειας αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν απέναντι στη βιομηχανία θα πρέπει να τους δίνουμε και πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πλαίσιο λειτουργίας να υπάρχει ασφάλεια κανονιστική ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κλάδος ε, του Χάλιβα απειλείται σαφέστατα και απειλείται και από το ντάμπινγκ, το ακούσαμε, αλλά όχι μόνο. Και από την παραγωγή χάλιβα ε, με χώρες που κάνουν εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και σας ζητώ κύριε Αντιπρόεδρε να δείχνετε μεγαλύτερη φιλοδοξία διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το βάρος της ε, βιομηχανίας και να μην ε, προστατεύουμε τη βαριά βιομηχανία. Παρακαλώ να πάρει μια απόφαση το Συμβούλιο και να βγάλετε και επίσημη αντακίνωση για μέτρα αντι-dumping για ε, ελάχιστη τιμή αγοράς για προστασία στα εξωτερικά σύνορα για να προστατευόμαστε από τις εισαγωγές ή τουλάχιστον να μειωθεί η τιμή της ενέργειας. Η χαλιβουργία ε, βαραίνει πάρα πολύ. 60.000 θέσεις εργασίας μόνο στην Ισπανία και 14 δισεκατομμύρια. Κυρίως στη, ε, ε, στην περιφέρεια που είναι σημαντική η χώρα των Βάσκων. Θα πρέπει αυτές οι κινήσεις να γίνουν αν γίνεται από αύριο το πρωί. Ο κύριος Δεμπάκερ, ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις από πλευράς μου. Ίσως θα μπορούσε να επεκταθεί ο Επίτροπος περισσότερο στις επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής για το ρίσκο και τον κίνδυνο των προϊόντων και των έργων που επιλέγεται. Σήμερα τα επιτόκια είναι σχεδόν αρνητικά, είναι ουσιαστικά μηδενικά. Άρα αυτό μπορεί να σημαίνει και μετατόπιση του κινδύνου στα έργα όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΦΣΥ επεμβαίνουν ενδεχομένω. Δεύτερη ερώτηση για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είπατε ότι τα δύο τρίτα των ε, έργων έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε να ξεφύγουμε από τη θεμελιώδη έρευνα και να πάμε σε πιο εφαρμοσμένη και πιο κοντά στην αγορά. Έχετε στοιχεία τα δύο τρίτα που πάνε στην έρευνα και ανάπτυξη Ποια είναι αυτά τα έργα όμως από τεχνολογική απόψεω είναι κοντά στην κυκλοφορία στην αγορά είναι θεμελιώδη έρευνα. Η κυρία Κίτσον darling, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για εσά, κύριε Επιτροπέ, Αντιπρόεδρε. Σε αντίθεση με τα όσα υπόθηκαν, εγώ καλωσορίζω το πρόγραμμα δράση για τη χαλιβουργία, το τελευταίο και το προηγούμενο, και εγώ αυτό θέλω να δω τώρα τη δράση, όχι μόνο το πρόγραμμα, να αρχίσει συγκεκριμένα να υλοποιείται. Και αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχικοί κρατών έχουν την ευκαιρία να λάβουν κάποιες αποφάσεις για αποφασιστική δράση. Συμφωνώ ότι στο Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε να κινούνται. Είδαμε μια σειρά ε, ε, ετών εμπλοκής και υπάρχουν κυβερνήσεις που συνεχίζουν να ε, μπλοκάρουν το χαμηλότερο τέλος, το lesser duty και αν το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίσει την τακτική του ε, θα ε, υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και είναι πραγματικά ηρωνικό, γιατί έχουν χάσει 6.000 θέσεις εργασίας και παραπάνω στη βόρειο-ανατολική Αγγλία, έχουμε πληγεί τα μάλα, είναι ολέθριο για την τοπική οικονομία και ταυτόχρονα, και εδώ είναι το ζήτημα, ταυτόχρονα που βλέπουμε ντάμπινγκ με φτηνό χάλιβα να μπαίνει, οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν μέτρα στη δική τους ε, ε, εισαγωγή ε, χάλιβα ψυχρής έλασης που έχει έρθει και έχει κατακλείσει όλη την αγορά. Άρα αυτά τα μέτρα ε, έχουν ε, αρθεί μόνο μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς θα βοηθήσετε το χάλιβα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάνουν οι Αμερικανοί με το δικό τους γιατί εμείς στο εργατικό κόμμα με τους συντρόφους αγωνιζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να πούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χαλιβουργία μας. Και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη βιομηχανία μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος eh, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα χαλιβουργία. Πριν από 20 χρόνια εγώ ήμουν επικεφαλής ε, μιας μικρής επιχείρησης επεξεργασίας χάλιβα και ε, τώρα ε, ετοιμάζεται να κλείσει και άλλες εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν με αποτέλεσμα τεράστια ανεργία. Μετά για τις διάφορες μορφές ενέργειας, τις ανανεώσιμες, ε, θα μπορούσε να μας πει ο Επίτροπος κάτι για το πρόγραμμα που βασίζεται στο υδρογόνο, η χρήση, για τη χρήση του υδρογόνου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης η Πολωνία έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί μετασχηματιστές υψηλής τάσης και η Τσεχική Δημοκρατία το σκέφτεται διότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να βελτιώσουμε το σύστημα διανομής της ενέργειας διασυνοριακά. Στη βιομηχανία πρέπει πομένουν να γίνουν μια σειρά πληρωμών ανακυλοβάτα, αναπόδοση και αυτό εισάγεται τώρα κάτι παρόμοιο στην Τσεχική Δημοκρατία. Καταφέραμε όμως να αναστείλουμε το έργο τελικά. Ε, τι πιστεύετε εσείς στην Κομισιόν γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Καλώ επιστρέψατε εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Κάποια σχόλια και μετά μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα σήμερα η Επιτροπή ε, μας παρουσιάζει σημαντικές κατευθύνες γραμμές για να σώσουμε τη χαλιβουργία. Δεύτερον, όσον αφορά την κυκλική οικονομία που είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κομισιόν φέτος, ξεκινήσαμε τη συζήτηση ε, σήμερα το πρωί. Είναι σημαντικό να θέσουμε στόχους ώστε να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείε για καινοτομίες και να τις ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσουν τα υλικά με νέους τρόπους. Χαιρόμαστε λοιπόν που ακούμε ότι εστιάζεται σε αυτό και στην Κομισιόν. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το περιβάλλον καινοτομία στην Ευρώπη. Δεν είμαστε αρκετά ανοιχτοί για νέε καινοτομίε. Αυτό ισχύει και για την συνεργατική οικονομία, το sharing economy. Ε, σε ορισμένες πόλεις απαγορεύεται το Airbnb, Uber, ε, η Κομισιόν έχει ξεκινήσει να δημιουργεί ένα νέο ε, ε, πλαίσιο για αυτή την sharing economy. Πώς πάνε τα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα αίτημα πρώτα απ' όλα και μια σκέψη μετά. Το αίτημα είναι το εξή, ε, κύριε Αντιπρόεδρε. Μπορείτε να μας στείλετε την παρουσίαση που μόλις κάνατε γιατί ακούσαμε πολλά νούμερα, πολλά δεδομένα, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Ήταν πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσουμε και να καταλάβουμε. Οπότε θα ήθελα να την έχω. Και αν μπορείτε να μας στείλετε και στοιχεία για τα όσα συμβαίνουν με την εύση. Μην μου πείτε ότι όλα βρίσκονται στο ίντερνετ γιατί όπω ξέρουμε Όλοι ναι υπάρχουν, αλλά θέλουμε και κάποια στοιχεία αξιολόγηση, γιατί εμεί είμαστε μία αρχή απολογισμού. Λαμβάνουμε αποφάσει, θέλουμε να βλέπουμε κατά πόσο οι αποφάσει μα κινούνται όντω προ την κατεύθυνση που θέλουμε. Οπότε κάποια αξιολόγηση. Τέλο πάντων, για να δούμε αν επιτυχάνουμε του στόχου μα. Τώρα, ε, για τα ερευνητικά έργα, ε, πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία διαφορετικά μετά από την επταετία μπορεί να έχουμε κάπου ε, ε, κατακαιρματιστεί μεταξύ έργων ε, σπαταλώντας χρήματα εδώ και εκεί. Χρειάζεται κάποια συγκέντρωση τώρα όσον αφορά την έρευνα και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί και πιο γενναιόδοροι. Πολλοί φτάνουν στο πρώτο βήμα και το περνάνε αλλά δεν περνούν το δεύτερο παρότι είναι άριστοι. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα να υπάρχει δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε έργα που έχουν αξιολογηθεί ως άριστα να, να ε, παραβλέπονται. Η κυρία Σπυράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθατε εδώ. Σήμερα διάβασα τη συνέντευξή σας στην εφημερίδα Λεκό και σύμφωνα με τη γαλλική έκδοση οι κυβέρνησεις παίζουν ρόλο αλλά το κυριότερο είναι στα χέρια των ιδιωτών επενδυτών. Στη χώρα μου, λόγω της κατάστασης των πραγμάτων, δεν υπάρχει κανένα ε, έργο από το ΕΦΣΙ που να χρηματοδοτείται στην Ελλάδα, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εσείς προτίθεστε να αρχίσετε μια εκστρατεία για την έλλειψη ε, ενημέρωσης για να ενθαρρύνεται μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ιδιώτες επενδυτές να χρηματοδοτηθούν από αυτό το ταμείο. Και δεύτερη ερώτηση αφορά τη συμπληρωματικότητα. Ε, πρόσφατα έχετε δημοσιεύσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις συμπληρωματικότητες μεταξύ ΕΦΣΥ και Ταμείο Συνοχής και τα Ταμεία τα διαρθρωτικά. αυτό θέλω να σας ρωτήσω, είναι κομμένο και ραμμένο για να χρησιμοποιηθεί για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Προσφύγων μάλλον, γιατί οι χώρες ε, αγγίζουν τα όρια τους ως προς τις δυνατότητες δράσης. Ευχαριστώ η κυρία Βέρνερ. Äh, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, και εγώ μερικά σχολεία για την Κίνα έχω. Ε, έχει μια επιθετική οικονομική εξάπλωση η Κίνα που πολλοί το θεωρούν μεγάλη απειλή, όχι μόνο για τη χαλιβουργία και όλες τις εξαγωγικές βιομηχανίες, φωτοβολταϊκά, ακόμα και σιδηρόδρομοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε τώρα και μπράβο τη και καλά έκανε, αλλά δεν θα πρέπει να αντιδρούμε, θα πρέπει και να δρούμε πρώτα απ' όλα. Ε, γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι χρειάζεται μια βιομηχανική στρατηγική που να ασχολείται και με το πώς θα διαφυλάξουμε την παραγωγή αξίας στην Ευρώπη και θέλω να σας ρωτήσω, θα υπάρξει ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική που να έχει και μια συνεκτική ε, βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και θα την εξασφαλίζει και αυτό το καλό στόχο το 20% θα το ξανανοίξετε. Έχω και μια ερώτηση συγκεκριμένη για τη χαλιβουργία. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κλάδος μπορεί να βγει από την κρίση ε, απλώς και μόνο αν σφίξετε αυτή τη μέγενη έχετε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσετε τον κλάδο να φύγει από αυτή τη μέγενη. Ευχαριστώ. Τζορίνιο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε. Είστε επίτροπος για την ανταγωνιστικότητα και για την απασχόληση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, δεν προσελκύουμε όμως τις αναγκαίες επενδύσεις και βιομηχανία κινδυνεύει. Όταν βλέπουμε τις τάσεις για τη χώρα μας που ανήκουν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη συνέπεια. Χρειαζόμαστε διεθνωτικές αλλαγέ στην ευρωπαϊκή οικονομία. χωρί αλλαγέ το δυναμικό των ευρωπαϊκών οικονομιών ποτέ δεν θα απελευθερωθεί και να διορθώσει τι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Υπάρχει ασυνέπεια όμω, όπω σα έλεγα στα μέτρα. Πολλές προτάσεις επιφέρουν, συνεπιφέρουν ανισορροπίες και παγιώνουν τις ανισορροπίες και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ε, φτώχειας αντί ένας θετικός κύκλος ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να, με τις συστάσεις που βλέπουμε δεν θα βρούμε τη λύση βράχη μεσοπρόθεσμα. Αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε σε ερωτήσεις και στα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Επίτροπο. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για τι ερωτήσεις. Νομίζω ότι λογικό θα ήταν να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις και απαντήσεις γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας πολλούς ευρωβουλευτέ. την κυρία Σπυράκη Φερρυπίν που βοηθούσε βοήθησε πάρα πολύ να περάσει ένα μήνυμα για το έργο του Ευρωπαϊκού Στατικικού Ταμείου. Τι είναι το ΕΦΣΥ, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς να συνδυάσουμε τους άλλους πόρους με τους πόρους του ΕΦΣΥ. Χρειαζόμαστε αγγελιοφόρους να διαδώσουν το μήνυμα σε όλες τις χώρες. Αλλά και στις περιφέρειες χρειαζόμαστε ανθρώπους έτσι. Αν δείτε τις χώρες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα το ΕΦΣΙ είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία. Ίσως και κάποιος άλλος. 22 χώρες χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ. Τι κάνουμε. Οι αντιπροσωπείες μας στις χώρες αυτές επιταχύνουν τις δραστηριότητες. Ο Μιγγέλ που κάθεται δίπλα μου, που εργάζεται στο γραφείο μου, πήγε στη Ρουμανία την περασμένη εβδομάδα να συζητήσει με τις αρχές, να τους εξηγήσει πώς το ΕΕΦΣΙ μπορεί να συνδυαστεί με άλλους ευρωπαϊκούς πόρους και συζήτησε και με τις τράπεζες. Αν δείτε τις γειτονικέ σας χώρες, τη Βουλγαρία, ήδη τέσσερις ιδιωτικές τράπεζες έχουν πάρει πόρους από το ΕΕΦΣΙ και θα χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτά τα χρήματα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Σε κάποιες χώρες υπάρχει έλλειψη, έλλειψη πώς να το πω, έμπνευσης ή βούλησης να υποβάλλουν προγράμματα. Ο ταχύτερο δρόμο να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι να πει κανεί στι τράπεζε. Αν θέλετε να εξυπηρετήσετε καλύτερα του πελάτε σα με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με χρηματοδότηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο. Οι ιδιωτικέ τράπεζε κάνουν τη δουλειά τα καταφέρνουν. Και βέβαια μετά χρειαζόμαστε και καλά προγράμματα συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Αυτές οι χώρες που ωφελήθηκαν περισσότερο είχαν κάποιους ανθρώπους που ενδιαφερόταν για τη χρήση του ΕΦΣΙ και διαβίβαζαν το μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. Άρα μας ωφελεί και εμάς να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να κινηθούν. Επισκέφτομαι τα κράτη-μέλη και δέχομαι και πολλούς ανθρώπους από διάφορες περιφέρειες και επανειλημμένα τους ε, εξηγώ πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Για το Χάλιβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Είπατε ότι πρέπει να θρήσουμε τις δυνάμεις μας και να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του πακέτου για τα αμυντικά εμπορικά μέτρα. Ελπίζω ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα θα διαβιβάσουν το μήνυμα στις αντίστοιχες κυβερνήσεις σας. Τώρα είναι η ώρα να αποτελματωθεί η κατάσταση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας στο παγκόσμιο εμπόριο. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια ότι το dumping και η μεγάλη προσφορά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Αν συγκρίνουμε την Αμερικανική βιομηχανία με την Ευρωπαϊκή, οι Αμερικανοί είναι πιο αποδοτικοί όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας. Και γι' αυτό έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη βιομηχανία μας να επενδύσει στο μέλλον της. Και πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις κυβερνήσεις μας να μειώσουν τη φορολόγηση της ενέργειας. Αν δείτε τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών, Υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση της ενέργειας ή τη τιμολόγηση της ενέργειας. Η ενεργειακή ενιαία αγορά ίσως μέσω μακροπρόθεσμα να βοηθήσει. Υπάρχουν όμως πολλά εθνικά μέτρα που θα πρέπει να δρομολογηθούν για να επικρατήσουν ίσες συνθήκες. Και η ρυθμιστική ασφάλεια, η σιγουριά αυτή που έθεσε ο κύριος Λεβαντόσκι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κατά την άποψή μου ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου είναι σημαντικότερος από το ΕΦΣΥ. Ο το πυλώνα τι σημαίνει. Προγράμμα ταινίας αγορά, αλλά και εντοπισμός των φραγμών για τις επενδύσεις που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Διότι υπάρχουν φραγμοί σε όλα τα κράτη-μέλη και βοηθάμε τα κράτη-μέλη να τα εντοπίσουν και να τα άρουν ένα-ένα. Η διαφορετική κατάσταση στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ από ό,τι σε εμά. Σε πολλά σημεία, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να αναφερθώ λεπτομερώς τώρα. Όχι μόνο ο χάλιβας, τα ίδια μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Να μην εστιαζόμεθα μόνο επί του χάλιβος, ας δούμε και το μέλλον της ενεργοβόρου βιομηχανίας, των ενεργοβόρων βιομηχανιών, διότι χρειαζόμαστε παραγωγή και τη βαριά βιομηχανία χρειαζόμαστε, παρόλο που προωθούμε ιδέες για την κυκλική οικονομία. Η κυρία Κάλλας ρώτησε. Πώς ξέρουμε ότι τα χρήματα δεν θα φερεθούν από την έρευνα και καινοτομία. Κανείς δεν μπορεί να το κηθεί. Πολύ συχνά είναι εύκολο να κόψει κανείς από την έρευνα την καινοτομία. Από έρευνα και ανάπτυξη αντί από άλλες υποδομές ή από άλλες δαπάνες. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι άειλο. Σε αυτή την επιτροπή πολλοί θα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που προβάλλουν τα κράτη-μέλη, είμαι σίγουρος. Το συ, ο συμβουλευτικός αυτός κόμβος λειτουργεί πολύ καλά. Έχουμε ήδη 90 αιτήματα και δύο τρίτα των αιτημάτων προέρχονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν συμβουλές. Πώς να χρησιμοποιούν πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή πώς να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων τους. Ο κόμβος αυτός φαίνεται ότι λειτουργεί αρκετά καλά, θα πρέπει να το προωθήσουμε. Λοιπόν, σε λίγες εβδομάδες θα ανοίξει και η πύλη για τα προγράμματα. Αυτή η πύλη του διαδικτύου ήρθε από τις ιδιωτικέ τράπεζες επενδυτικές. Είπαν ότι μπορούν επενδύσουν περισσότερες, ε, περισσότερα χρήματα σε, σε ιδιωτικά προγράμματα υποδομές και είπαν ε, γιατί δεν φτιάχνετε εμεί το σελίδα για να υποβάλλονται περισσότερα προγράμματα. Υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων. Για να υποβάλλουν εκεί τα προγράμματα και τι προτάσει. Και σε λίγε εβδομάδε θα ανοίξει αυτή η πύλη του ιστοτόπου και θα χρησιμοποιήσουμε για χρήματα για διαφήμιση σε διάφορα περιοδικά και στο σελίδε που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό κόσμο. Και χρειαζόμαστε και εδώ τη βοήθειά σα. Όταν δείτε ότι λειτουργεί, περάστε το μήνυμα στι περιφέρειέ σα, στου δήμου, στι κυβερνήσει, στον ιδιωτικό τομέα Πείτε τους, αν θέλετε καλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ εκείνων που χρηματοδοτούν τα προγράμματά σας, στέλνετε τα προγράμματά σας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα. Και όταν ανοίξει, περάστε το μήνυμα και διαδώστε το μήνυμα. Πείτε ότι είναι καθετικό. Ο πολλαπλασιαστής είναι περίπου 17 από πλευράς μικρομεσαίων είναι πολύ ψηλότερος. Ο πολλαπλασιαστής από πλευράς προγραμμάτων είναι χαμηλότερος. Ε, εξαρτάται βέβαια από την ζήτηση εξαρτάται και από την ποιότητα των ε, προγραμμάτων βλέπετε. Λοιπόν, έρευνα και ανάπτυξη ορίζων 2020, επενδύσεις. Είμαι πεπισμένος ότι 2,2 δις από τον ορίζοντα 2020 στον ΕΦΣΥ θα ωφελήσει πολύ περισσότερη έρευνα από τα 2,2 δις. Βέβαια, αν τα 2,2 χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελιώδη πανεπιστημιακή έρευνα, τότε θα ήταν 2,2 για τη βασική έρευνα. Τώρα τα χρήματα χρησιμοποιούνται για πιο εφαρμοσμένη έρευνα που έχει κατέθει στην αγορά. Αληθεύει αυτό. Όλοι το ξέραμε ότι θα συμβεί. Λοιπόν, ε, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος της χρηματοδοτήσεως για την ε, καινοτομία είναι μεγαλύτερος. Υπάρχουν θετικές πτυχές και αρνητικές πτυχές ανάλογα με το πώς βλέπει κανείς τα πράγματα και τι θεωρεί πιο σημαντικό. ETS, υπάρχει μια πρόταση, ξέρετε, το εμπόριο αυτό του ε, ρήπων το ETS με το εμπόριο σχετίζονται. Όσο πιο πολύ παραγωγή έχουμε εδώ, τόσο πιο καλό το κλίμα. Και το ETS ε, ε, επιβάλλει ισότιμες συνθήκες, το σύστημα εμπορίας ρήπων. Λοιπόν. Μπορούμε ποικιλοτρόπως να το δημιουργήσουμε, το οικοδομήσουμε το ETS. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς εκτός του χάλιβα που ανταγωνίζονται και καθορίζονται τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όπως ε, κεραμικός τομέας, ε, χαρτοπολτός, χαρτοβιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να συμβιβαστούμε και είναι στα χέρια τα δικά σας και του Συμβουλίου να αποφασίσετε ποιος είναι ο κατάλληλος συμβιβασμός. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε υπεύθυνο συμβιβασμό. Δηλαδή ένα βρύ φάσμα βαρέων ε, βιομηχανιών θα παραμείνει στην ε, Ευρώπη. Τώρα, βιωσιμότητα των προγραμμάτων και των έργων ήταν ένα άλλο θέμα που ετέθη. Δεν έχω πολλά να πω για την ποιότητα συγκεκριμένων μεμονωμένων προγραμμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα έχει επιλέξει. Υποσχεθήκαμε και τηρήσαμε την υπόσχεσή μας να μην παρέμβουμε στην επιλογή των προγραμμάτων. Ο πίνακας βαθμολόγησης δείχνει μία εικόνα στην Επιτροπή Επιλογής για να κάνει τις επιλογές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αργότερα θα μας ενημερώσει, θα υποβάλει εκθέσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αυτής και θα προβεί σε διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων και της ποιότητας των προγραμμάτων. Είναι πρόημο τώρα να τοποθετηθώ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα ξεχωριστά προγράμματα. Γεωγραφική δικαιοσύνη τώρα. Οι μεγαλύτεροι χρήστες ή δικαιούχοι του ΕΦΣΙ είναι η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θυμάμαι με ποια σειρά. Και όπως σας είπα, 22 κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν το ΕΦΣΙ, αλλά υπάρχουν και χώρες με προβλήματα. Γι' αυτό εκείνος και εγώ και άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όλοι μαζί παρακολουθούμε, βοηθάμε τα κράτη-μέλη και επαναλαμβάνω αυτά που είπα. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Εάν θέλετε η πληροφορία θα σας δώσουμε ό,τι θέλετε. Χρησιμοποιήστε τις αντιπροσωπίες μας στα κράτη-μέλη σας. Οργανώστε εκδηλώσεις για ε, επιχειρηματίες, ε, για επενδυτές, ανθρώπους των τραπεζών, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Στην Ελλάδα, Φερρυπίν, χαίρομαι που έχουμε αυξήσει την παρουσία μα εκεί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έστειλε περισσότερου ανθρώπου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να βοηθήσει τι αρχέ να βρουν προγράμματα και να τα χρηματοδοτήσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ο ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να στεστούμε επί του ιδιωτικού τομέα περισσότερο από τι κυβερνήσει. Στην Ελλάδα, Φερρυπίν. Συνάντησα πολλούς βιομηχάνους και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και κάθε φορά ακούνε για πρώτη φορά ότι δεν χρειάζονται την έγκριση της κυβερνήσεως αν θέλουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Κάθε φορά είναι νέα μαντάτα για αυτούς όταν τους συναντώ. Άρα πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά, να ενημερωθούν. Ιστοσελίδα, έχουμε έξοχη σελίδα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και το ΕΦΣΥ και βρίσκεται κάθε πρόγραμμα εκεί στην ιστοσελίδα. Και όταν διαφημίζω το ΕΦΣΥ χρησιμοποίησα αυτά τα προγράμματα, διότι έτσι ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Βλέπουν οι μεν τι έκαναν οι δε. Οι πλατφόρμες τώρα. Υπάρχουν δύο-τρεις πλατφόρμες και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, θετικά μάλλον προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αν είχα χρόνο θα εξηγούσα περισσότερο ε, τις πλατφόρμες, τι είδους πλατφόρμες διαθέτουμε. Ε, προσπάθησα να μεγιστοποιήσω τον αριθμό πλατφορμών ή να έχω όσο το δυνατόν περισσότερε πλατφόρμε για να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ για μικρότερα προγράμματα ομαδοποιώντα. Τώρα, συνεργασίε για τα οικονομικά θέματα. Θα παρουσιάσουμε κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ ισχύουν οι κανόνε ε, τη Ευρωπαϊκή Ενώση για τη συνεργατική ε, οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι στη σωστή πλευρά, να η ιστορία να δείξει ότι έκανα σωστές κινήσεις. Και αυτή η συνεταιριστική οικονομία μπαίνει στην αγορά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο κανονισμό που δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια και αντιβαίνει στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα σύγχρονα αυτά μοντέλα, τα επιχειρηματικά, ποιο θέλουμε να εξασφαλίσουμε, την ανάπτυξη, την νέα ανάπτυξη, τον καινούριο κόσμο ή το παλιό ρυθμιστικό βαρύ περιβάλλον. Γι' αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να σκεφτούν αν θα ήταν λογικό να αλλάξουν κάποιους κανόνες που σκοτώνουν τις νέες επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και για ευκαιρίες. Και τέλος, νομισματική πολιτική και, και εικόνα του κινδύνου. Οπότε ε, ε, ε, σωστή δανειοδότηση, η σωστή νομισματική πολιτική μειώνει τον κίνδυνο όσον αφορά τη δανειοδότηση. Αυτά έχω να πω σε αυτό το μέτωπο. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και αν έχετε άλλες ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε επιθυμείτε στείλτε μου ένα μήνυμα ή μπορούμε να συναντηθούμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την οριζόντια προσέγγιση. Το ίδιο έκαναν και τα μέλη μας όπως αντιληφθήκατε. Θέλουμε να συζητάμε τα πάντα μαζί σας, όχι μόνο το ΕΦΣΥ, που είναι ίσως το πιο σημαντικό, αλλά και την απλούστευση για τη χαλιβουργία, των οριζόντα 2020, το ETS, το πρόβλημα της Κίνας, τις ε, νέες οικονομίες αγοράς, ε, της ΕΙΠΑ, τον ανταγωνισμό και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να ξανασυναντηθούμε, διότι δεν έχουμε τελειώσει το σκληρό μας έργο. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για τη συζήτηση. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 8 διακυβέρνηση της ενία αγοράς. Ποιο είναι το ζήτημα εδώ, να διευκολύνουμε τη ζωή των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Συναρπαστικό θέμα. Να κάνουμε τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες να λειτουργούν ευκολότερα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Hello. Hello. Easy, easy life is not easy question. Easy life for, for our business and industries. Λοιπόν, να διευκολύνουμε τη ζωή επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Ε, η, την παρουσίαση θα μας κάνει η Διευθύντρια Βαλεντίνα Σουπέρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεθνής Ανάπτυξη φυσικά, διότι όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, για επενδύσεις, για την ανταγωνιστικότητα και για μεγάλη ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οπότε θα μιλάμε για όλα αυτά, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσά ε, και σε όλους σας ε, αξιότιμα μέλη. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρισκόμαι εδώ σήμερα, ειδικότερα μετά από την ομιλία ενό τόσο ε, υψηλού επίπεδου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στι προσδοκίε σα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Λέγομαι Βαλεντίνα Σουπέρτη, διευθύντρια ε, πόρων στην DG Grow για... και ασχολούμαι και με αυτά τα ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς και ε, η Λοράνς Δερισμόν δίπλα μου είναι η αρμόδια ε, τμήματάρχης. Γιατί είναι τόσο μεγάλη μου χαρά σήμερα η παρουσία μου εδώ. Ακριβώς για όλα αυτά που μόλις είπατε κύριε Πρόεδρε. Αφενός ε, είναι ε, σημαντικό η ενιαία αγορά που είναι η κινητήρια μηχανή για την πρόθεση των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη να λειτουργεί αποτελεσματικά ε, σε όλα τα επίπεδα και με εύκολο τρόπο. Είναι ωραίο στα λόγια αλλά δύσκολο στην εφαρμογή. Ωστόσο, και αυτό θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα, και θα θέλαμε την υποστήριξή σα ουσιαστικά για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα, αυτά τα εργαλεία και την ενημέρωση. Είναι ότι σήμερα λοιπόν αυτό που θέλω να πω, σήμερα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία σειρά εργαλείων τα οποία εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό, το να διευκολύνουμε τις ζωές των επιχειρήσεων ε, και να τονίσω ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Τι λέμε εδώ τώρα, για να είμαι σαφής δεν λέμε τα κλασικά στοιχεία, ε, νομοθετικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς. Δεν μιλάμε για ε, την οδηγία για τις ε, ιατρικές συσκευέ. Δεν μιλάμε για όλα αυτά τα πολυάριθμα νομοθετήματα που γνωρίζουμε όλοι μας. Ούτε μιλάμε για διαδικασίες επιβολής του νόμου. Δεν μιλάμε δηλαδή για επίσημες διαδικασίες που ενδέχεται ε, να ξεκινήσει η Κομισιόν σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, ε, της διαδικασίας παραβάσης όπως λέμε. Εδώ αντιθέτως μιλάμε για πρακτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ώστε να λειτουργεί ενιαία αγορά στην πρακτική. Λοιπόν, δεν θέλω να με βαρεθείτε, οπότε πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω τα εργαλεία αυτά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ενιαία αγορά και πώς εφαρμόζεται στην Ευρώπη και τα σχετικά εργαλεία. Έχουμε το Europe Advice που παρέχει πληροφορίες σε απλή γλώσσα, σε πολλές γλώσσες, σε όλους τους πολίτες χωρί ορολογία και υπογραμμίζω ξανά στι μικρέ επιχειρήσει, γιατί οι μικρέ επιχειρήσει είναι αυτέ που δεν έχουν τα μέσα να γνωρίζουν του κανόνε, δεν, δεν έχουν τα λεφτά για να πληρώσουν δικηγόρου. Οπότε εμεί προσφέρουμε αυτό το εργαλείο παροχή απλών και περιεκτικών πληροφοριών για την ενιαία αγορά σε αυτέ. Στη συνέχεια Μιλάμε για σύνδεση μεταξύ και επαφή μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της Κομισιόν κατά την υλοποίηση της νομοθεσίας. Τι είναι αυτό? Ονομάζεται EIMI. Ε, είναι σύστημα διαχείρισης πληροφοριών. Είναι η βάση δεδομένων μας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 10 νομοθετημάτων, την οδηγία πεσπασμένων εργαζομένων, την οδηγία υπηρεσιών, την οδηγία επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και άλλα ε, που περιμένουν στην ουρά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο πληροφορικής που εξυπηρετεί το σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των άρμοδιων αρχών των κρατών μελών με στόχο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τρίτον, κάτι που μάλλον σας είναι γνωστό, αλλιώς ε, αυτή είναι η μέρα μου, το Solvit. Τι είναι το Solvit. Είναι ένας μηχανισμός, ένα δίκτυο μεταξύ κρατών μελών, αρχών κρατών μελών και της Επιτροπής με στόχο να γίνεται μια προσπάθεια επίλυσης ε, διαφορών όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή σε θέματα ε, νομοθεσίας ενίας αγοράς. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί, λαμβάνουμε καταγγελίες μέσω του Solvit και μεριμνούμε ώστε να γίνουν οι επαφές μεταξύ ας πούμε της Πολωνίας και της Γερμανίας, απλά δίνω ένα παράδειγμα, ώστε και οι δύο αρχές να μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα μεταξύ τους. Χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε επίσημες διαδικασίες. Γιατί είναι ελκυστικό αυτό το σύστημα, διότι είναι ένας άτυπος μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Τέταρτον, ε, μιλάμε για τον πίνακα βαθμολόγησης. Ε, ε, αυτός είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου έχουμε μια συγκριτική επισκόπηση των επιδόσεων των κρατών μελών σε θέματα κανονών της ενιαίας αγοράς. Έτσι γνωρίζουμε ποιος θα πάει καλά, ποιος λιγότερο καλά από τα κράτη-μέλη σε θέματα ενιαίας αγοράς. Λοιπόν, θα είμαι σύντομη γιατί θα ακολουθήσει και η προβολή ενό βίντεο που θα σας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα από μένα και με εικόνες με πιο παραστατικό τρόπο θα σας παρουσιάσει αυτά τα εργαλεία αλλά το πρώτο μήνυμα προς εσάς είναι το εξής εμείς στην Κομισιόν γνωρίζουμε και τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν ότι τα εργαλεία αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά λειτουργούν μια χαρά ωστόσο πρέπει να γίνουν περισσότερο γνωστά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Διότι ελπίζουμε ότι εσείς με τις πολλές επαφές που έχετε στις εκλογικές σας περιφέρειες θα διαδώσετε αυτή την πληροφορία ε, ύπαρξης αυτών των εργαλείων. Επίσης, επιτρέψτε μου να σας υπογραμμίσω ότι τα εργαλεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όσον αφορά πρωτοβουλίες σημαντικές της Κομισιόν όπως ε, η στρατηγική της ενιαίας αγοράς. Γιατί ιδιωτηρισμένα από αυτά τα εργαλεία ενδέχεται να αποδειχθούν ωφέλιμα όταν αναφερόμαστε ας πούμε στην ε, ε, ψηφιακή ενιαία πύλη που είναι μια ενιαία πύλη για όλα τα θέματα που αφορούν την ενιαία αγορά και την οποία προετοιμάζει τώρα η Κομισιόν και για το Solvit. Το Solvit ε, παρεμπιπτόντως από μόνο του ήδη αναφέρεται στη στρατηγική της ενιαίας αγοράς, επίσης αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας ε, στα τέλη του περασμένου έτους. Οπότε η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ είναι η βελτίωση και η περαιτέρω ενίσχυση του Solvit ως ενός ε, εύκολου τρόπου προώθησης της ενιαίας αγοράς και διασφάλισης της σωστή λειτουργίας ε, πρακτικά της ενιαίας αγοράς χωρίς να περνούμε από περίπλοκες και μακροχρονίες ε, και δαπανηρές διαδικασίες. Θα κλείσω εδώ και αν δεν διαφωνείτε μπορούμε να δείξουμε τώρα το βίντεο και μετά αν έχετε ερωτήσεις ευχαρίστως να προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. και παρακαλούμε βοηθήστε μας να διαθώσουμε το νέο. Ευχαριστούμε. Αξιότιμη κυρία, λοιπόν, ας δούμε τώρα το, την ταινία αυτή που ονομάζεται Spectacle. Europeans go to another EU country every year to find a better job, to study in university, to do business, or to spend a well-earned holiday. A lack of information, incorrect application of an EU rule, or simply a misunderstanding can make life difficult.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 Thank you very much. That's all. That's all. Αυτό ήταν όλο. Ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση, να ακούσουμε ερωτήσεις, σχόλια. Anybody would like to say something. Uh, Συνάδελφε Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Ναι, έχω να πω κάποια πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε καλύτερα με τους πολίτες θα ήθελα να ξέρω, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από τα κοινωνικά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσα hits υπάρχουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα των πολιτών, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε σε ποιες χώρες δεν χρησιμοποιείται, όπου υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Στη ΣΤΟΑ ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα ε, και ονομάζεται Σιλό και στρατηγική για τους σωλήνες. Πώς οι κυψέλες γνώσεις επικοινωνούν στην Ευρώπη. Τα Σιλό της γνώσης ε, που είναι η νέα αντίληψη. Συνάδελφε Κούλιτσεκ, σας ευχαριστώ. Έχω την εξής ερώτηση. Πολύ συχνά παραπονιέται ο κόσμος Όσον αφορά το διοικητικό άχθος, θεωρούν ότι είναι υπερβολικό το άχθος. Έχετε λάβει κάποια μέτρα λοιπόν για να μειώσετε αυτό το άχθος, το διοικητικό άχθος, το βάρος αυτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Κάλτε. Ευχαριστώ πολύ. Κέλλη, συγγνώμη. Έλεγα επί καιρό ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι χειρότερα, οι χειρότεροι φορείς όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις στον κόσμο. Διότι κάνουμε πολλή δουλειά και μας επικρίνουν τα μάλα. Και δεν δίνουμε απαντήσεις στις περισσότερες επικρίσεις ή οι απαντήσεις όταν δίδονται δεν προβάλλονται και βασιζόμαστε μόνο στον εαυτό μας για να διβάσουμε το μήνυμα. Και γι' αυτό καλωσορίζω όλος ιδιαίτερος το υπέροχο αυτό την ταινιούλα που είδαμε που δείχνει αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα περισσότερα από αυτά. Μου άρεσε η αναφορά στο Solvit, βλέποντας τα συνολικά στοιχεία, βοηθά πολλούς το Solvit. Πόσοι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξή του, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διβάσουμε το μήνυμα. Είναι καλό το να ετοιμάσει κανείς ένα βίντεο, αλλά άλλο αυτό και άλλο να μάθει ο κόσμος γι' αυτό. Πώς μπορείτε να οικοδομήσετε σε αυτή την πολύ καλή βάση που δημιουργήσατε για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, να τους δείξουμε ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Να μην μαθαίνουν μόνο τα ΜΜΕ τι γίνεται, που πολύ συχνά ε, παρουσιάζουν φανταστικά στοιχεία, μια φανταστική εικόνα για τον Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την πραγματική. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, άλλος που ζητά το λόγο. Πιο γενική ερώτηση έχω εγώ. Ε, ο Επίτροπος ο κ. Μπαρνιέ πριν κάποια χρόνια, πριν 7 χρόνια, ξεκίνησε τη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είχε τους 12 άθρους της ευρωπαϊκής αγοράς που ήθελε να πετύχει. Στόμα μας είναι η διακυβέρνηση, η εργαλεία στην ενία αγορά. Δεν αναφερόμαστε στις μεταρρυθμίσεις εντός των κρατών μελών, αλλά στην ενιαία αγορά. Και ο κ. Μπαρνιέ, ο επίτροπος ο κ. Μπαρνιέ, είχε αναλάβει 12 σκοπούς, αν θέλετε. Ποιο τομέα, ποιο στοιχείο από τα σημείο από τα 12 σας ενδιαφέρει στην έκθεσή σας. Πνευματικά δικαιώματα, Φερρυπίν. Πολλά διαφορετικά θέματα αναφερόταν. Όταν τελείωσε τη θητεία του, Θέλουμε να ξέρουμε ποια ήταν η αποτίμηση. Ερώτηση, πού βρισκόμαστε όσον αφορά τους 12 σκοπούς, άθλους, στόχους για την ενιαία αγορά, για την υλοποίηση ενιαίας αγοράς. Πριν από 7 χρόνια βρήκαμε 150 κενά περίπου στην ενιαία αγορά. Εσείς πώς τα βλέπετε, τα κενά που υπάρχουν. αναφέρονται επιχειρήσεις, η βιομηχανία και να διευκολυνθούν, να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη. Περί αυτού πρόκειται. Ίσως μπορούμε να βρούμε απάντηση μετά αν είναι περίπλοκη ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις και με τα σχόλια. Όλα αυτά δείχνουν ε, ότι το θέμα είναι πράγματι και ενδιαφέρον και σημαντικό. Παρεμπιπτόντως ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Με ακούτε καλά. Ωραία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Όσον αφορά τα νούμερα, σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την ερώτηση. Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα εργαλεία αυτά ε, είναι ιδιαίτερα επιτυχή. Και μπορώ να σας δώσω στοιχεία, να σας στείλω μετά από τη συνάντηση αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία. Να σας πω για παράδειγμα ότι για το Your Europe ε, είχαμε 22.000 ερωτήματα το 2015, ότι το Solvit χειρίστηκε πάνω από 2.200 περιπτώσεις, ότι το EMI επέτρεψε πάνω από 10.000 ανταλλαγές πληροφοριών. Τα νούμερα υπάρχουν. Και αυτό δείχνει τη γενικότερη επιτυχία των εργαλείων αυτών. Πιο συγκεκριμένα δείχνει ότι όταν οι χρήστες και οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν, το ποσοστό ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ο δείκτης ικανοποίησης και αυτή είναι η αφετηρία μας. Δεδομένων αυτών, και αυτό τώρα σχετίζεται και με τη δική σας ερώτηση. Ε, τότε η προκλήση, μάλλον οι προκλήσεις είναι οι εξής. Ε, οι βασικές δύο ε, προκλήσεις είναι ότι ναι πρώτον ναι τα εργαλεία είναι επιτυχή όταν είναι γνωστά. Το θέμα όμως είναι πώς οι πολίτες στην Ευρώπη γνωρίζουν τα εργαλεία αυτά. Και ας είμαστε ειλικρινείς τώρα με τους εαυτούς μας ε, και πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Ακούστηκε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο ότι ε, το Solvit δεν είναι τόσο γνωστό. Ε, και μέσω αυτού του βίντεο, αλλά ξέρετε εμεί όταν σα δείχνουμε ένα τέτοιο βίντεο σε μια σημαντική επιτροπή του Κοινοβουλίου δεν είναι παρά ένα στοιχείο, μία από τι πολλέ δράσεις που σχεδιάζουμε για την ε, ευαισθητοποίηση. Έχουμε ήδη επισκεφθεί την Επιτροπή ΙΜΚΟ, την Επιτροπή Γιούρι, τώρα βρισκόμαστε εδώ και όσους περισσότερους επισκεφθούμε τόσο πιο ικανοποιημένοι θα είμαστε γιατί έτσι θα επέρθει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα δεν είναι για εσάς ή για εσάς ε, προσωπικά κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη είναι ότι όλοι εσείς θα μπορέσετε να διαδώσετε τις πληροφορίες Ωστόσο εργαζόμαστε εντατικά εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνουμε, προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την ενημέρωση του εξωτερικού κόσμου όσον αφορά αυτά τα εργαλεία. Προσπαθούμε να σκεφτούμε πιο σύγχρονα, πιο... Ε, ε, μπορούμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διότι ξέρετε... Ε, πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ενημερώνεται μόνο μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωσης, οπότε προσφέρουν πολλέ δυνατότητε και μετά υπάρχει και μια, υπήρξε και μια ερώτηση για το θέμα του άχθους και της απλούστευσης. Τι θέλει λοιπόν αυτό το θέμα της απλούστευσης και της ε, συγκέντρωση όλων των εργαλείων που έχουμε ώστε να δίνουμε ένα πιο απλό, ευθύ μήνυμα, κατανοητό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Όλα αυτά σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την εμβληματική πρωτοβουλία της Κομισιόν στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίας αγοράς αλλά και με τη στρατηγική ενίας αγοράς Το ανέφερε και η Επίτροπο Βιανκόφσκα όταν ήρθε εδώ για να εξηγήσει τα διάφορα, τις διάφορες εργασίες. Λοιπόν, πρώτον, η ψηφιακή ενιαία απειλή. Ξέρετε ότι ετοιμάζουμε μια πρόταση τώρα. Βέβαια το θέμα βγαίνει εκτός των όριων της παρουσίασής μου εδώ, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά μελετάμε αυτή την πρόταση που θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι η ενημέρωση προς πολίτες και επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το σημείο πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων ε, στα διάφορα εργαλεία θα είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και πιο εύχριστα. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης, ένα single entry point για θέματα ενιαίας αγοράς. Οπότε ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απάντησα τώρα και μερικώς για το θέμα του διοικητικού άκθου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ε, μετά με τα όσα ρώτησε ο κύριος Ρίμπιχ και ευχαριστώ που το θίξατε διότι τώρα ξεκινάμε το θέμα αυτό ε, αφορά μια πιο στρατηγική χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουμε μια πιο οργανωμένη χρήση γιατί ουσιαστικά μέσω των εργαλείων αυτών εμείς συλλέγουμε πληροφορίες. Μπορούμε να παρατηρούμε τι γίνεται, να κάνουμε συγκρίσεις και να αποκομίζουμε διδάγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για το Solvit, αυτός ο μηχανισμός άτυπης επίλυσης διαφορών αποτελεί κομμάτι των τροχών εργασιών, όχι μόνο για να λειτουργεί μόνος του. Και τέλος, έχουμε ξεκινήσει τώρα να εξάγουμε ε, πληροφορίες από τις διάφορες ανταλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο Solvit ώστε να αποκομίσουμε πιο συστημικά διδάγματα ειδικότερα όσον αφορά τις ε, υποθέσεις που ονομάζουμε δομικής σημασίας ε, δομικής σημασίας όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτά ε, ε, μπορώ να σας πω προς το παρόν τώρα. Λοιπόν, ε, κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, κύριε Μπούζεκ, αναφερθήκατε στην πράξη νέας αγοράς και στις 12 δράσεις. Μου έχουν πει ότι οι δύο δράσεις από τις 12 έχουν επιτευχθεί. Τώρα προτεραιότητα έχει η υλοποίηση της ε, στρατηγικής ενιαίας αγοράς. Πράγματι, γιατί, γιατί ο Επιτρόπος Μπαρνιέ ξεκίνησε το έργο του τότε, ήταν αρμόδιος για την ενιαία αγορά, ενώ ο Ταγιάννη ήταν υπεύθυνο για την ε, ε, βιομηχανία, ξεκίνησε πράγματι την πράξη ενιαίας αγοράς και τις σχετικές προτάσεις, αλλά μετά, ειδικότερα μετά από την ε, συγχώνευση του πρώην κομματιού της εσωτερικής αγοράς με το κομμάτι της βιομηχανίας στο ίδιο χαρτοφυλάκια στη νέα επιτροπή του Γιούνκερ. Το σημαντικό έγγραφο πολιτικής ε, που θα βοηθήσει να επιτύχουμε την ενιαία αγορά είναι η στρατηγική για την ενιαία αγορά. Αυτό το έγγραφο πιστεύω πρέπει να θεωρούμε ότι είναι τώρα το έγγραφο αναφοράς ε, σε θέματα πολιτικής. Όπως είπε ε, και η Επιτροπός Μπιανκόφσκα σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, τρεις είναι οι βασικοί στόχοι για να εμβαθύνουμε ή να πετύχουμε καλύτερα την ενιαία αγορά. Πρώτος είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η δεύτερη είναι ο εξυγχρονισμός των οικονομιών και της βιομηχανίας ειδικότερα. Αυτό αποτελεί κομμάτι τη στρατηγική ενίας αγορά. Αλλά τρίτο, πολύ σημαντικό που σχετίζεται με τα όσα είπαμε σήμερα εδώ, είναι η επιτόπου εφαρμογή, η πρακτική εφαρμογή. Ελπίζω να απάντησα επαρκώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια. Σήμερα Έχουμε επαφές με την ε, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Digi Growth, με τον πιο άμεσο τρόπο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για τις απαντήσεις σας, για την παρουσίαση. για να διευκολύνετε τη ζωή των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. και εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην υπηρεσία σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και που ε, έχετε το χρόνο να συζητήσετε μαζί, μαζί μας και είμαστε στη διάθεσή σας όποτε το θελήσετε. Ευχαριστώ να πάτε στο καλό. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα. Μελέτη με θέμα βιομηχανία 4.0. Παρουσίαση από το Γιάννη Σμιτ, από το κέντρο ε, των υπηρεσιών για στρατηγική και αξιολόγηση. Σας ενημερώνω ότι τη μελέτη αυτή την ανέθεσαν το 2015 συντονιστές στη Ήτρε με στόχο να δούμε ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια επιτυχή βιομηχανία 4.0. Ε, Στο δημόσιο τομέα να δούμε τι μέτρα πρέπει να ε, ληφθούν και τι βήματα πρέπει να γίνουν. Πολλά ακούμε για τη βιομηχανία 4.0, 4.0. Ξέρουμε ότι είναι το μέλλον μας και θα θέλαμε να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα από τον κύριο Γιάνν Σμιτ. Κύριε Διευθυντά, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα, πού βρισκόμαστε και τι μελιγενέστε. Τι σημαίνουν όλα αυτά και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε από πλευράς της βιομηχανίας 4.0 γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε οι πάντα ηγέτες και πρωτοπόροι σε αυτά τα θέματα αλίμονο. Έχετε αμέσως τον λόγο, παρακαλώ. Hello, can you hear me? Yes, certainly we can hear everything. Βεβαίως. Ε, μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Έχω μια παρουσίαση PowerPoint, αν θέλετε να ανοίξετε το σύστημα. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για την παρουσίασή μας, οπότε um, θα είμαι σύντομος και ελπίζω συνεκτικός για να έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις και απαντήσεις στη συνέχεια. Έχετε και την έκθεση σε γραπτό κείμενο με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι μπορούμε εμείς να πούμε σήμερα προφορικά. Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης, ε, της παρουσίασης. Είναι πραγματικά να ενημερώσουμε για την πολιτική αυτή που μας ζητήσατε, τι είναι η βιομηχανία 4.0, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος, ποιες ε, είναι οι βασικές αγορές, τι γίνεται με την τεχνολογική αλλαγή. Και πολύ σημαντικά είναι τα η τεχνολογική, η κοινωνική αλλαγή και η αλλαγή στο υπόδειγμα το επιχειρηματικό. Αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτή τη βιομηχανία 4 σε αυτά τα θέματα. Okay, στο βαθμό που μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Και τέλος με μια αξιολόγηση και ε, συστάσεις για την πολιτική. Λοιπόν, οι σημερινοί στόχοι να μπορούμε να ενημερώσουμε τη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική, ποιο δρόμο να ακολουθήσει στο μέλλον, να εστιάσουμε στην σύνδεση μεταξύ των ψηφιακών τεχνολογιών και των βιομηχανικών προϊόντων και ε, υπηρεσιών. Ακούσαμε και προηγουμένως πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ατζέντα. Να δούμε λοιπόν τι συγκεκριμένη ε, βιομηχανία, τι σημαίνει η βιομηχανία 4.0 και τι επιπτώσεις έχει τεχνολογικές, κοινωνικές και αλλαγές, όπως είπαμε στο υπόδειγμα των επιχειρήσεων. Η βιομηχανική πολιτική έχει αναλυθεί το τελευταίο διάστημα, 60-70 χρόνια. Έχει περάσει από διάφορα στάδια, ε, από τη δεκαετία του 70 που χαρακτηριζόταν από επιλεκτικούς στόχους ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους και πολλές φορές δεν ε, θεωρήθηκε πάρα πολύ επιτυχημένη. Στη συνέχεια η πολιτική αφορούσε ε, ε, το ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιομηχανία και από το 2000 είχαμε νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Τα στοιχεία στην έκθεσή μας δείχνουν και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα μερίδια της βιομηχανίας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας στα διάφορα κράτη-μέλη και ε, διαφέρουν ε, από χώρα σε χώρα. Τι είναι λοιπόν η βιομηχανία 4.0? Είναι η οργάνωση της παραγωγής που βασίζεται ε, σε συσκευές που επικοινωνούν αυτόματα κατά τη διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής. Βασικά είναι συστήματα με κομπιούτερ ε, που παίρνουν αποφάσεις γιατί μεμούνται την πραγματικότητα σε μια εικονική πραγματικότητα και ελέγχουν τις φυσικές διαδικασίες. Εδώ χρειάζονται κάποια προπετούμενα για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Μεταξύ αυτών είναι η ανάπτυξη ε, συμπεφωνημένων προδιαγραφών, αλλαγές στις ε, μεθόδους εργασίας και στην οργάνωση, ε, χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της ηλεκτρονικής διεύθυνση. Ε, διαθεσιμότητα εργαζομένων, έρευνα, κατάρτιση, ε, επαγγελματική ε, εξέλιξη και το νομοθετικό νομικό περιβάλλον. Ένα μεγάλο πεδίο και σχετιζόμενοι όροι είναι το ίντερνετ των αντικειμένων, το ίντερνετ των υπηρεσιών και το βιομηχανικό ίντερνετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ αυτών. Ποια είναι η στρατηγική για να είμαστε ηγέτες στην αγορά. Αυτό το είδαμε στην αρχική ε, ε τεκμηρίωση. Συντονίζουμε τις, ε, τη ζήτηση για να οδηγηθούν ε, οι κλάδοι στην καινοτομία μέσω δικτύωσης μεταξύ των εταιριών και συνεργασία ε, των κλάδων. Ωραία είναι το λες αυτό, αλλά πρέπει και να εφαρμοστεί. Σημαίνει ψηφιακή ολοκληρώση σε διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, σε κύκλους προϊόντων, κύκλους ζωής ε, και μια σειρά άλλα ε, που έχουν να κάνουν με την παραγωγή κάποιων προϊόντων. Το θέμα είναι και είναι μεγάλη πρόκληση πώς θα ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλα αυτά τα δίκτυα αξιών. Η στρατηγική ηγετική θέση στην αγορά συνδέεται και με τη στρατηγική ε, προσφοράς, έτσι μια διπλή στρατηγική. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι αυτό από μέσα. Πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν αυτά τα προβλήματα και τις προκλήσεις, αλλά λίγες λέγουν και ιδιαίτερα λίγες μικρομεσαίες ότι είναι έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Και διαφέρουν και οι απόψεις στη βιομηχανία και ε, στους ερευνητές στο ποιο βαθμό επηρεάζονται και άλλοι τομείς. Ε, δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ούτε απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Είναι μεγάλα τα προβλήματα, το κόστος και οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή ασφάλεια, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ε, προσωπικών δεδομένων, ιδιωτική σφαίρα, λειτουργικότητα των συστημάτων, προστασία περιβάλλοντο, ασφάλεια και υγιεινή. Για το πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Και το κόστος αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων αυξάνεται όσο περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Διάφορα δημόσια ιδρυμάτα θεσμοί δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη σε πολλέ χώρε για να βελτιωθεί η ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο ε, στο διαδίκτυο και αυτό αυξάνει και το κόστος βέβαια. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη ευρεία κλίμακα για έρευνα σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης από απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Um, Ποια είναι η κοινωνική αλλαγή. Αν δούμε την κοινωνία στο σύνολό τη, δεν έχει πάρει είδηση. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, δεν είναι ευνοϊκά διακείμενες αυτό από ότι πιο μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες. Τα συνδικάτα παραμένουν επιφυλακτικά και έχουν ε, πολλές αφιβολίες και επιφυλάξεις και υπάρχει ένα έλλειμμα προθυμίας να προσαρμοστούν στην ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως ακούσατε και προηγουμένως, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο χάσμα δεξιοτήτων. υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 θα χρειαστούν 825.000 ειδικοί για την ψηφιακή πραγματικότητα που μας λείπουν. Και ε, τα τεχνικά και άλλα προαπαιτούμενα και προσόντα είναι πολύ ψηλότερα στον νέο αυτό κόσμο. Και ε, θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους εργασίας για να προσαρμοστούμε στην βιομηχανία 4 και να έχουμε και συντονισμένες προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Είναι άνηση η προσφορά τέτοιων δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσόντων και αναμένεται να αυξηθεί. Με τη μετανάστευση όμως μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό για να δούμε πώς αλλάζει το επιχειρηματικό υπόδειγμα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγάλα τα προβλήματα και τα, ε, οι προκλήσεις, το κόστος, ο κίνδυνος, μειωμένη ευελιξία και στρατηγική ανεξαρτησία. Στη Γερμανία έχει γίνει μια έρευνα σε ένα δείγμα χιλίων επιχειρήσεων με ένα τζίρο 500.000 έως 125 εκατομμύρια και έδειξε ότι και 35% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν παίζουν σημαντικό ρόλο έως καθόλου οι ψηφιακέ τεχνολογίες. Το βασικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να μένουν ανταγωνιστικές. Και για τις μικρότερες εταιρείες αυτό το ποσοστό ήταν 52% των εταιριών αυτό. Θα πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή βιομηχανία να παραμείνει ανταγωνιστική με άλλα μέρη του κόσμου, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα κτλ. Ε, συνολική αξιολόγηση λοιπόν και εκτίμηση. Η βιομηχανία 4 ε, ε, έχει πολύ περισσότερα ενδεχόμενα ωφέλη για τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά συνδέεται και με μεγαλύτερο κόστο, κίνδυνο και απειλέ. Θα υπάρξουν νικητέ και ειτημένοι και τα επόμενα 10-15 χρόνια θα χρειαστούν για να προσαρμοστούμε τι σημαίνει αυτό για την πολιτική και τις συστάσεις. Σίγουρα αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή και πρωτοβολίε υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθούν να έχουν επιτυχία και θα πρέπει βεβαίω να συνεχιστεί αυτή. Ωστόσο τα μεμονωμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκτιμήσουν την θέση της πολιτικής τους για να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της δικής τους οικονομίας και βιομηχανίας και στους στόχους. Υπάρχουν βασικά ελλείμματα και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε για την πολιτική αυτή, η βιομηχανική η πολιτική δεν είναι πάντα συντονισμένη γύρω από ένα συντονισμένο στόχο για την βιομηχανία 4 ή το βιομηχανικό διαδίκτυο είναι κατακαιρματισμένο και πολύ σημαντικό εστιάζεται ε, στην τεχνική έρευνα και ε, παραμελεί τον ανθρώπινο παράδειγμα, τα social κοινωνικά, social, δηλαδή τα κοινωνικοτεχνικά συγγνώμη και άλλα στοιχεία. Ελπίζω να μην ε, στραπατσάρισα πάρα πολύ το θέμα τρέχοντας όσο πολύ από τις διαφάνειες. Είναι ένα βρύ πεδίο που πρέπει να καλυφθεί. Ήθελα να σας πω αυτά τα σημεία και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και με τον συνάδελφό μου. Thank you very much uh, for your... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω και την ε, έντυπη εκδοχή, μπορείτε να τη βρείτε. Είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο. Uh, για να τη μελετήσουν όλοι. Όλα μπροστά στα μάτια μας είναι. Κύριε Κόλλιτσεκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αυτός είναι ο στόχος του βιομηχανικού κόσμου για το μέλλον. Όμως, είναι ένα θέμα επίμαχο. Συζητείτε. Το συζητούν θεωρητικοί, επαΐοντες. Και στον τρίτο κόσμο έχουμε την έναρξη της εκβιομηχάνησης. Όμως όλοι συμφωνούν σε κάτι. Θα υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι με το κατάλληλο, ε, κατάλληλη εκπαίδευση, υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης και πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ελοχεύει. Μας περιμένει στη γωνία, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και θα έπρεπε να είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διαφορετικά, αυτό το μόρφωμα των 28 κρατών μελών δεν έχει καμία πιθανότητα να επιβιώσει. Βέβαια, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για την κατάσταση αυτή. Εξίσου σημαντικό είναι να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει οι πολίτες. Δεν είναι και όλοι πανέξυπνοι με IQ 130 για να γίνουν ερευνητές. Ούτε όλοι είναι αρκετά επιδέξιοι για να μπορούν να εργαστούν σαν μηχανικός, σαν τεχνικός σε κέντρα ρομποτικής. Δεν είναι όλοι σε αυτή τη θέση, δεν έχουν όλοι αυτού του είδους τα προσόντα. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως εκ τούτου είναι να ε, μπορέσουμε να δώσουμε καλές λογικές θέσεις απασχόλησης σε εκατομμύρια ανθρώπους, εργαζομένους όλα θα αυτοματοποιηθούν και όσο αυτοματοποιούμεθα τόσο πιο πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να βρουν κάποια θέση στην αγορά εργασίας. Δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά στην έρευνα, στην ανάπτυξη και σε άλλους τομείς που χρειάζονται πολλά προσόντα. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που προκύπτει από όλα αυτά. Υπάρχει ένα νέο επίπεδο εκβιομηχάνησης όχι μόνο μετακίνηση της βιομηχανίας προς χώρες που έχουν πιο χαμηλό εργατικό κόστος και χαμηλότερες περιγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, αυτό το συζητάσαμε πριν και εκτενώς, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και άλλη απειλή. Να χάσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η απειλή που ελοχεύει. Βλέπουμε ότι πολλές χώρες έχουν ξεπεράσει την Ευρώπη τεχνολογικά. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόιερ έχει το λόγο. Κυρία Τόγια μάλλον, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχασα το πρώτο μέρος, αλλά θα τη διαβάσω πολύ προσεκτικά. Η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα τόσο που έχουμε προετοιμάσει μια κρόση αύριο ε, αλλά τελικά θα αντικατασταθεί από αυτό του σχεδιασμού της ενέργειας που είναι πιο επίγον. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό σίγουρα. Μια ερώτηση που θέλω να κάνω από τις πολλές είναι Έχω μελετήσει αυτά που γράφουν διάφοροι εμπειρογνώμονες, προβλέψεις για το μέλλον και κάτι που απογραμμίζεται διαρκώς είναι ότι θα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο πολλών επιχειρήσεων και ότι πολλές επιχειρήσεις από ε, κατασκευαστές προϊόντων θα γίνουν παραγωγή υπηρεσιών ταυτόχρονα. Ε, ε καθώς θα βάλουμε την αυτοματοποίηση για παράδειγμα σε αυτό το βιομηχανίες είναι θεωρητικές αυτές οι προβλέψεις ή πραγματικά μεταλλάσσονται έτσι σιγά σιγά οι επιχειρήσεις ε, από προϊόντα δηλαδή θα παράγουν και προϊόντα και υπηρεσίες αλλάζοντας φύση και τι θα κάνουμε, εσείς λέτε ότι θέλετε να αφήσετε να εξελιχθεί η αγορά χωρίς πολλές παρεμβάσεις, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι όταν θα ζητηθεί προσωπικό εξειδικευμένο, καταρτισμένο με συγκεκριμένο τρόπο, με πολλαπλές δεξιότητες, διότι ναι, θα έχουμε μία μείωση της απασχόλησης, αλλά μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση για νέες δουλειές Υπάρχουν ε, κάτι που γίνεται ε, όσον αφορά την εκπαίδευση ε, στον τομέα αυτό από εμά, από τα πανεπιστήμια, από τον βιομηχανικό τομέα. Τι άποψη έχετε εσεί. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κάπαλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, κύριε Σμιτ για αυτή την εμπεριστατωμένη μελέτη για τη βιομηχανία 4.0. Τα μεγαλύτερα θέματα που μας απασχολούν εδώ για την ψηφιοποίηση έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Γίνεται και πολλά και υπάρχει λόγος. Ε, γι' αυτό παρακαλέσαμε και σας αναθέσαμε να κάνετε αυτή τη μελέτη, να μοιραστείτε μαζί μας την πραγματογνωμοσύνη σας. Αναφερθήκατε σε τρεις διαστάσεις που έχουν σημασία για την αλλαγή, δηλαδή η τεχνολογική αλλαγή, η κοινωνική αλλαγή και ε, οικονομική αλλαγή, ε, αλλαγή οικονομικού υποδείγματος. Μας είπατε πώς βλέπετε τη τεχνολογική αλλαγή με πολύ πρακτικό τρόπο. Χθες άρχισε η έκθεση Τσέμπιτ ε, που έχει να κάνει με ε, το διαδίκτυο των αντικειμένων, το iCloud και τέτοια πράγματα που κανονικά αφορούν τους πάντες. Και φτάνουμε και ε, στην κοινωνική αλλαγή εδώ. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν καν τι σημαίνει βιομηχανία 4.0. Το λέτε και στη μελέτη, είναι πάρα πολύ τεχνικός όρος και χρησιμοποιήθηκε για να δώσει ιδιαίτερη πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση ε, της γερμανικής μικρομεσαίας ε, ε, βιομηχανίας και πραγματικότητας. Το είπατε και εσείς σήμερα όμως αφορά και τη ζωή και την εργασία των περισσότερων ανθρώπων. Πραγματικά είναι κοινωνική αλλαγή και αυτή η κοινωνική αλλαγή βεβαίως έχει και νέες απαιτήσει που φέρνει και στον κόσμο της εργασίας και τις δεξιότητες και τα προσόντα που περιμένουμε από τον κόσμο. Ε, με αυτή την ψηφιακή αλλαγή λοιπόν και την τεχνολογική αλλαγή θα πρέπει να μπορούν να συμβαδίζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό χρειάζεται η προσαρμογή. Ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό εδώ στην Ευρώπη. Πάνω από 400 δισεκατομμύρια έχει υπολογιστεί στην Ευρώπη εάν η εσωτερική αγορά η ψηφιακή ολοκληρωθεί. και δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι τεχνολογία τεχνολογίες καινοτομίας και τεχνολογίας καλπάζει από ότι γνωστή και παραδοσιακή κλάδη της οικονομίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε, να έρθουμε πιο κοντά. Και είπατε ότι το 35% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν ότι δεν τους αφορά η ψηφιοποίηση. Άκουσαν, άκουσαν. Αυτό λέει και μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διείσδυση των μικρομεσαίων ε, στο επιγραμμικό εμπόριο. Είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ είναι τεράστιο το δυναμικό. Γι' αυτό χρειάζονται και οι πλατφόρμες αυτές που αναφέρεται στη μελέτη. Έχω μια συγκεκριμένη όμως ερώτηση εγώ, διευκρινιστική έχετε επισυνάψει ε, μια ε, συγκεκριμένη μελέτη ε, για μια περίπτωση που μελετήσατε αριθμό 5 για την Κίνα και εδώ αναφέρετε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Κίνας, το Internet Plus και το Made in China. Γνωρίζετε ότι το, η Κινέζικη Βουλή, το Λαϊκό Κογκρέσο, αποφάσισε ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα και η Κίνα θέλει να δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας αλλού στις υπηρεσίες, θα τις καταργήσει από τις κλασικές ε, βιομηχανίες και πώς το βλέπετε αυτό το Made in China και το Internet Plus που προσανατολίζεται να φύγει από την παραγωγή αγαθών για να παράγει ε, υπηρεσίες και ψηφιοποιημένα. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Sorry. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Να σας κάνω μια σύντομη ερώτηση. Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε τις διαφορές ε, από την άψη της βιομηχανίας ρομποτικής. Τις διαφορές λοιπόν μεταξύ της δικής μας Υπήρου και των πολιτείων της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Χονγκ Κόνγκ, Ταϊβάν, Σιγκαπούρης. Πού βρισκόμαστε γενικώ. Γενική ερώτηση. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Σε σύγκριση με την παγκόσμια οικονομία. Είμαστε μπροστά όπως και στην πολιτική για το κλίμα. Έχετε το λόγο. Oh, Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πολύ εύστοχες. Και φυσικά υπάρχουν περιορισμοί για το τι μπορούμε να μιλήσουμε και να συμπεριλάβουμε σε μια έκθεση. Πολλοί κόσμοι μιλάει για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν έχω τέτοια άποψη κατά πόσο είναι ή όχι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η ετικέτα ή κάποια ονομασία. Πάντως σίγουρα κάτι συμβαίνει. Αν θέλει κανείς να το δει από την άψη των βιομηχανικών επαναστάσεων, κάτι πολύ ενδιαφέρον που υποστηρίζουν όσοι υποστηρίζουν αυτή την έννοια κάθε φορά που γίνεται μια βιομηχανική επανάσταση αλλάζουν οι ηγέτιδες βιομηχανίες ε, αλλάζουν, ε, αλλάζει το μέρος όπου βρίσκονται οπότε αν βρισκόμαστε σε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα αλλάξει ε, η βιομηχανική κυρίαρχη του κόσμου σε σχέση με το παρελθόν δεν ξέρω αλλιώς θα ήξερα που να βάλω τα λεφτά μου αν Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, συζητείται πολύ. Ουσιαστικά τα πάντα κινούνται γύρω από τα βασικά σημεία που ανέφεραν και εδώ οι ευρωβουλευτές κατά ερωτήσεις. Είναι ότι για να παίξει ένας πολίτης το παιχνίδι του Industry 4.0 ε, χρειάζεται πολλές γνώσεις και εξειδίκευση. Και πώς αποκτά κανείς αυτές τις γνώσεις, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Ε, αν δούμε τα, η βιβλιογραφία που έχει εκπονηθεί στην Γερμανία, το ζήτημα δεν είναι μόνο περισσότερες δεξιότητες, είναι αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τρόπου σκέψης. Κάτι που το καθιστά μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Για παραδείγμα, το ιδανικό προφίλ ε, για την πρόσληψη ενός ατόμου σε μια επιχείρηση φαίνεται να είναι κάποιος που έχει διδακτορικό σε ε, υπολογιστικές επιστήμες και που μπορεί να λειτουργήσει ως προσωπικός ψυχολόγος και σύμβουλος, ένας διαχειριστής ε, επικοινωνιών, ε, διαχειριστής διαπροσωπικών σχέσεων, ικανός να έχει ευρεία εικόνα του μέλλοντος της βιομηχανίας και επίσης ικανός να συμμετάσχει σε μια συνεργασία μεταξύ συνδικάτων και επιχειρήσεων ώστε όλοι να συνεργάζονται αρμονικά. Έτσι, ξέρετε, οδηγούμαστε μερικές φορές να σκεφτούμε ότι κάποια ε, από τα ζητήματα που συζητάμε για τη βιομηχανία ίσως είναι λίγο τοπικά. Διότι δεν μπορεί κανείς να κάνει όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα, σίγουρα όχι ένα άτομο. Παρότι λοιπόν χρειαζόμαστε εξειδίκευση και ε, ε, εξειδικευμένες ικανότητες για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ακόμα παραπάνω μάλιστα. Ε, ο, ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κάποια όρια στο τι μπορεί να κάνει και στο πόσο μπροστά μπορεί να κινηθεί μαζικά όλη η βιομηχανία παρασύρτητας μαζί στην οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Είναι λίγοι αυτοί που σε υψηλό επίπεδο θα μπορούσαν, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχουν προκλήσεις για τους ε, ειδικού ε, στους υπολογιστές. Οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν είναι τόσο απλό να επιτύχουν τέτοια πράγματα. Κάποιοι λοιπόν θα αποκλειστούν από όλο αυτό λόγω έλλειψης δεξιοτήτων. Το έχουμε ήδη δει. Απλά για να ολοκληρώσουμε την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, και εκεί παρατηρούνται ελλείψεις. Παρότι το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται είναι χαμηλό, αν δείτε την έκθεση, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ε, ε, γεμίζει ξαφνικά με ανθρώπους από την Ινδία και το Βιετνάμ και άλλα μέρη του κόσμου, την Ινδονησία, ώστε να συμπληρώσουμε τα έχουμε εδώ τα κέντρα όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, στα κέντρα όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση όπως η Γερμανία αυτές οι χώρες ε, αντλούν ανθρώπους και από άλλα μέρη της Ευρώπης. Υπάρχει τεράστια δίψα για ανθρώπους με εξειδικευμένες ε, τέτοιες γνώσεις. Όσοι δεν έχουν τέτοιες δεξιότητες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες ε, στο μέλλον. Η όλη επίδραση για την απασχόληση έχουν γίνει κάποιες μελέτες, είναι περίπλοκο θα εξαρτηθεί από τον τομέα, από το μέρος του κόσμου, από τη χώρα. Η κάθε χώρα θα επηρεαστεί διαφορετικά. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, αλλά όλα είναι υποθετικά προς το παρόν. Αλλά όλα συγκλίνουν στην άψη ότι μάλλον θα αυξηθεί η απασχόληση, όχι πολύ, αλλά ότι κάθε ομάδα ε, ανθρώπων θα επηρεαστεί διαφορετικά. Είναι δύσκολο να δούμε αυτή τη στιγμή καθαρά το μέλλον της βιομηχανίας στο σύνολό της. Ωστόσο, έχει τεθεί το ερώτημα μεταξύ ε, στα συνδικάτων για το τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν έχουν τις γνώσεις και τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, ανταποκριθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία συγκεκριμένα το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει πραγματοποιήσει μελέτες επί του ζητήματος Ακόμα και αν βρούμε πολλούς εξειδικευμένους ανθρώπους ε, που έχουν τις δεξιότητες και αλλάξει μετά η οικονομία, τι θα κάνουμε με αυτούς μετά από 20-30 χρόνια αν εμφανιστεί κάτι άλλο. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι τεχνολογικά είναι απερχιωμένοι. Τώρα για τα ερωτήματα που αφορούν τυχόν μελλοντικέ αλλαγέ των επιχειρηματικών μοντέλων. δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αλλάξουν όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι αδύνατον. Αν αναλογιστείτε τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει βιομηχανία, φανταστείτε με μονομένες επιχειρήσεις να ενσωματώνουν τεχνολογίες στα συστήματα παραγωγής, στην ε, αλυσίδα αξίας, ε, να μοιράζονται ε, στοιχεία. Ελάχιστες μπορούν. Αυτό απαιτεί επενδύσεις, οπότε υπάρχουν βεβαιότητες για το θέμα αυτό αβεβαιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί με συγκεκριμένους προμηθευτές, θα γίνει να πάει κάτι λάθο. Ε, είναι και μεγάλο το κόστος των επενδύσεων αυτών, μερικές φορές υπερβολικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε δεν ξέρουμε αν αυτό είναι καλή πρόταση. Όλα αυτά με λίγα λόγια περιορίζουν την έκταση στην οποία το Industry 4.0 θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε όλου του τομείς της οικονομίας. Σε ορισμένου τομεί απλά δεν πρόκειται να πιάσει. Στην παρουσία φάση πιστεύω πρέπει να πούμε και το εξή. Κάτι που δεν ανέλησα εντό τη παρουσίαση, αλλά είναι σημαντικό, είναι η διαφορά του τι εννοώ εγώ όταν λέω Industry 4 και τι εννοούν άλλοι άνθρωποι όταν μιλούν για διαδίκτυο των ε, ε, πραγμάτων, των υπηρεσιών κτλ. Το Industry 4.0 αφορά την παραγωγή ε, βιομηχανιών. Είναι μια πολύ εστιασμένη δραστηριότητα από την αρχή της. Η βασική ιδέα ήταν η προετοιμασία της ε, γερμανικής παραγωγικής βιομηχανίας για το μέλλον. Αυτή η βιομηχανία είναι η πιο σημαντική, φυσικά η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε παρακολουθούμε ε, τι συμβαίνει εκεί. Και το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία, οπότε ε, πιθανότατα να μην, να μην τύχει τη ίδια προσοχή σε αυτέ τι χώρε του Industry 4.0. Τώρα για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια δεν αφορά μόνο τη μεταποιητική βιομηχανία αλλά και άλλες βιομηχανίες. Και μετά έχουμε και το διαδίκτυο των υπηρεσιών που φέρνει και τις υπηρεσίες ε, στο παιχνίδι του διαδικτύου. Εγώ σύστηκα πιστεύω ότι η έννοια του βιομηχανικού διαδικτύου της General Electric είναι αρκετά χρήσιμη διότι το βιομηχανικό διαδίκτυο ουσιαστικά περιλαμβάνει οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην οικονομία το οποίο μπορεί να μπει στο ίντερνετ, ε, να διαδικτυωθεί αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ε, συστήματα φωτισμού σε αστικές περιοχές, ε, σπίτια, οικοδομές, οικοδόμηση φραγμάτων, όχι απλά την μεταποίηση. Οπότε πρέπει να δούμε σε τι ακριβώς μιλάμε, αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το διαδίκτυο των πραγμάτων και για το βιομηχανικό διαδίκτυο. Στο Industry 4.0 ουσιαστικά αναφέρομαι μόνο σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Αλλάζουν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αρχίζουν να αλλάζουν το μοντέλο αρχίζει να πιάνει στις βιομηχανίες αυτές όπου αυτό είναι εφικτό. Αλλά ακόμη και μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών όπως είναι η Γερμανία, ε, εκεί θα σας πω ότι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο το Industry 4 θα αναπτυχθεί μέσα στην επόμενη 15 ετία, 20 ετία ίσως μέχρι να αρχίσει να χρησιμοποιείται ε, παντού ε, πέραν αυτών που αναπτύσσουν την ιδέα αυτή τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή θα δούμε πόσο πολύ έχει εξαπλωθεί. Αλλά ήδη από τώρα καλό είναι να προβλέψουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε θέματα όπως η απασχόληση. Η εκπαίδευση διαφόρων ανθρώπων είναι ενδιαφέρον ζήτημα επίσης. Είχαμε και το έγγραφο των όσων το σχεδίασαν όλο αυτό το Industry 4 λένε ότι απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγή συνεπώς του τρόπου διδασκαλίας διότι ουσιαστικά παίρνουμε ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί κλασικά σε πληροφορική, σε εξαγωγές, στον προγραμματισμό, ή σε υπολογιστέ ε, υπάρχει ένα στερεότυπο. Συχνά μα λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω, νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται μπροστά σαν υπολογιστή ατελείωτε ώρε και ενδεχομένω βγαίνουν έξω για να φάνε μια πίτσα και μετά ξαναγυρνάνε σπίτι τους στη δουλειά τους. Έτσι νομίζουμε ότι μοιάζει ένας προγραμματιστής υπολογιστή αλλά το Industry 4.0 πρέπει να μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, να ε, στέλνει ιδέες σε άλλες ε, βιομηχανίες, να υπάρχει κάποια ανταλλαγή, πρέπει να κατανοούν λοιπόν και επιχειρηματικές διαδικασίες, τις πολιτικές συνομιλίες με άλλες επιχειρήσεις ή άλλους πελάτες. Απαιτεί δηλαδή μια πλήρη μεταλλαγή της νοοτροπίας και της εκπαίδευσης. Κάτι που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί. Yes. Αυτό πρέπει να υποστηριχθεί η έννοιας του Industry 4. Μαζί και με άλλους πολλούς τεχνολογικούς παράγοντες. Uh, λοιπόν, νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Πάω στην τελευταία ερώτηση Ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε συγκρίση με άλλες χώρες. Επί του παρόντος δεν θα πρέπει να μιλάμε για Ευρώπη τώρα. Σε σύγκριση έχουμε και μεγάλα τμήματα εντός Ευρώπης. Η Γερμανία ηγείται εντός Ευρώπης. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Και οι πιο μεγάλες ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι η θέση με τους Αμερικανούς, κάποιους από τους Κινέζους ε, και τις πρώτες εταιρείες σε άλλες χώρες. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι στην πρώτη θέση με άλλες μεγάλες από άλλες χώρες. Εξέτασα κάπως άλλες χώρες όπως η Κίνα. Κάθε φορά που αυξάνονται οι μισθοί στην Κίνα θέλει η κινέζικη βιομηχανία να αυξήσει το τεχνολογικό επίπεδο και να συναγωνίσει σε υψηλότερο επίπεδο με τις βιομηχανίες τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Υπήρχαν κάποιες βασικές ερωτήσεις που δεν ετέθησαν. Ασφάλεια δεδομένων, αλλά τις ερωτήσεις των παρισταμένων πιστεύω τις απάντησα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πληρέστατη και ενδελεχέστατη απάντηση κάλυψε όλες τις ερωτήσεις μας. Στην επόμενη έκθεση ίσως μπορούμε να καλύψουμε και άλλα θέματα. Τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας και την ομάδα σας ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί σας. Ήταν το το τμήμα έρευνας που ήταν έλαβε αυτό του Ευρωκοινοβουλίου θέσαμε επιτάπητος ερωτήσεις. Χρειάστηκε χρόνος για τις απαντήσεις. Πρέπει να περιμένουμε και για την απάντηση του αντίστοιχου τμήματος ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ εκ νέου για την έκθεσή σας, για την παρουσίασή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση στις 9 το πρωί TTIP διαπραγματεύσει του TTIP 9 το πρωί πρωί πρωί στις 10 το πρωί ψηφοφορία και το υπόλοιπο πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι τις 12.30 αύριο τα πάντα στις 3 ακρόαση mm σημαντικότατη ακρόαση. Όλα μπροστά μας τα έχουμε. Για τους περισσότερους από εσά είναι το τέλος συνεδριάσεως διημέρης, αλλά για κάποιους από εσά πρέπει να περιμένετε λεπτά, λεπτά, έξι λεπτά, σε λεπτά και κλεισμένων των θυρών θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ο κύριος κύριε Κόλιτσεκ, σας ευχαριστούμε. Ξεκινήσατε με υπέροχο τρόπο το πρωί από ό,τι άκουσα, απουσίαζα, αλλά ήσασταν δραστήριος όλο το πρωινό, χρειαζόταν βλέπετε. Ο προκάτοχός σας ήταν, πώς να το πω, πολύ παλιό μέλος της Επιτροπής Ήτρο, ο κύριος Λάμστορφ και πολύ δραστήριος Ελπίζω λοιπόν να τον αντικαταστήσετε επάξια. Θα δούμε στο μέλλον. Είναι οι πρώτες μέρες. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Σε πέντε λεπτά θα συναντηθούμε ξανά με τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ.